Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Οι υπουργοί Ντάισελμπλουμ και Κάζιμιρ θα έρθουν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου που δίνουν. Περιμένουμε και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, αλλά καλύτερα να αρχίσουμε γιατί μέχρι τις 9 πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους Υπουργούς Οικονομικών που δέχτηκαν να λάβουν μέρος σε αυτή τη δημόσια κρόαση. Μάλιστα, έχουμε δημόσια κρόαση με 7 υπουργού από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Μάλτα σπάνια ευκαιρία ε, για συζήτηση με 7 ε, υπουργού Οικονομικών για τις δυνατότητες και τις επιλογές της δυνα... τις που μας δίνει μια δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης ε, και ποιες θα είναι οι συνέπειες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Η καθιέρωση της δημοσιονομικής ικανότητας ε, αναφέρεται ως πρόταση και στην έκθεση των πέντε προέδρων και από πολλούς ε, εμπειρογνώμονε ως πρόταση θεωρείται ως αναπόσπαστο τμήμα μιας ε, εύρυθμα λειτουργούσα οικονομικής και νομισματικής ένωσης και οι επιτροπές εκών και προϋπολογισμών απεξεργάζονται σχετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας με το θέμα αυτό της δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωζώνης. Και μάλιστα έχετε λάβει τα σχέδια έκθεσης ε, των συνεισηγητών Μπέγκε και Μπέρες με τη σαφή προσδιορισμό των πιθανών λειτουργιών και των βασικών πυλώνων της δημοσιονομικής ικανότητας. Κυρίως η πρόθεση της σύγκλησης ε, και η χορήγηση κινήτρων για τις μεταρρυθμίσεις, η απορρόφηση των ασύμετρων και συμμετρικών κραδασμών και το καθεξής. Και μάλιστα πρόσφατα το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο ε, δημοσίευσε ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο με ανάλυση των διαφόρων σενάριων και εναλλακτικών. Βέβαια, η συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολιτική συζήτηση και μεγάλη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με υπουργού οικονομικών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα. Και εκ μέρους του Ζαν Αρτουή, του Πρόεδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως Δίνοντα το λόγο, εκτό και αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Συμπρόεδρος. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου, ε, την ε, χαρά μου για αυτή την ε, συνεδρίαση που την περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο για το πέρας της ιδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό για να συναντήσουμε τους υπουργούς οικονομικών και να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό και της αξιολόγησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, της αναθεώρησης της ενδιάμεσης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Περβάνς περέ εκ μέρου και των δύο εισηγητών. Μαζί με τον Ράιμερ Μπέγκε και με το σύνολο της διαπραγματευτικής ομάδας ευχαριστούμε ειλικρινά του Υπουργού Οικονομικών που είναι εδώ μαζί μας. Είναι μια συνήθι περίσταση, αλλά νομίζω το θέμα του προπολογισμού της Ευρωζώνης είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και σας ευχαριστώ που απαντήσατε καταφατικά στην πρόσκλησή μας. Δεν θέλω να κάνω μακροσκελής παρεμβάσεις. Αυτό που θέλω είναι να σας ακούσω κυρίως εσάς και να δω μαζί σας πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό που σας προσφέρουμε, δηλαδή μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της, του προπολογισμού της Ευρωζώνης. Είναι ένα θέμα που είναι επιτάπητος. Πριν από την έκθεση Ντελόρ, μάλιστα. Η κρίση μας έδειξε ότι αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία για μια έκθεση για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης, από την αρχή ξέραμε ότι το θέμα αυτό θα τυθόταν στο τελευταίο τρίμηνο αυτής της χρονιάς, ανεξάρτητα από την έκβαση του Βρετανικού Δημοψηφίσματος. Και πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια. Ό,τι και να κάνετε εσείς, ε, γύρω από άλλα θέματα, όσο ενέργεια και αν ξοδέψετε για να τα αντιμετωπίσετε, αυτό το θέμα είναι αναπόφευκτο. Φαντάζομαι στη Σύνοδο Κορυφή στην Σλάβα θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε του προβληματισμού σα. Αλλά νομίζω ότι η υιοθέτηση αυτή τη έκθεση, τον Οκτώβριο κανονικά περιμένουμε να συμβεί του 2016, θα αποτελέσει μια βάση για εσά για να ξεκινήσει η συζήτηση στο εσωτερικό σας και να ετοιμάσετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του τέλους του 2016, ούτως ώστε να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την έκθεση των πέντε προέδρων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για να τη θέσουμε σε εφαρμογή, πιστεύουμε, μετά και να περιμένουμε όλες τις εθνικές εκλογές. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, μετά από την α ή τη β, τις α ή β εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε έτοιμοι από τώρα. Επίσης, στην έκθεση των πέντε προέδρων αναλάβα μια συγκεκριμένη δέσμευση και καλό θα ήταν να πάρετε συγκεκριμένη θέση. Τον ε, μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Γιατί στην έκθεση των πέντε προέδρων προβλέπεται ότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα ενσωματωθεί στην κοινοτική μέθοδο. Και αυτό θα έχει πολλέ συνέπειε. Και καλό θα ήταν βεβαίω να ακούσουμε τη γνώμη σας για όλα αυτά. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά το πρωτόκολλο που προβλέπει ε, με αλφαβητική σειρά να δώσουμε το λόγο στους υπουργούς ε, και στον Άρτη Ευχθέντα Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προηγείται ο Μισελ Σαπέν γιατί είναι σίγμα. Δεν κατάλαβα <laughs> τίποτα από αυτά που είπατε για το πρωτόκολλο. Εν πάση περιπτώσει, αλλά κάποιο πρέπει να κάνει το βάπτισμα του πυρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και του συμπροέδρου και του ευρωβουλευτέ. είναι η πρώτη φορά που έρχομαι ενώπιον σα, αλλά κάθε φορά έρχομαι με ιδιαίτερη χαρά. Και μάλιστα αν έτσι πραγματοποιούμε και το όνειρο του ε, Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ακόμη καλύτερα. Δεν έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιούμε συχνά τέτοια όνειρα. Και μάλιστα εσείς ε, προηγηθήκατε στο αξίωμα ε, του Υπουργού Οικονομικών και με διαδεχθήκατε κιόλα, οπότε ακόμη καλύτερα να μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε αυτό το όνειρο στις ε, εξαιρετικές προσπάθειες ε, των δύο συνεισηγητών, όπως είδαμε και από την παρουσίαση που μας έκανε η κυρία Μπερμάς Πέρες, ε, πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι καθόλου καινούριο. Είναι τόσο παλιό όσο και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το μόνο θέμα είναι ότι μόνο η ο νομισματικός πυλώνας ε, τέθηκε σε εφαρμογή με πολύ σχολαστικό και ακριβή τρόπο, κάτι που ήταν απαραίτητο φυσικά ε, για να θεσπιστεί, ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις λειτουργίες της, την ανεξαρτησία της και την ε, αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των νομισματικών θεμάτων. Αλλά μένει το οικονομικό σκέλος, ο οικονομικός πυλώνας και ο δημοσιονομικός που έμειναν μετέωρα. Οπότε έχουμε ένα μηχανισμό που δεν είναι και πολύ ε, ισορροπημένος. Και μάλιστα οι ανισορροπίες ε, φαίνονται όταν ε, ταρακουνιέται το κτίσμα και το βλέπουμε αυτό από την έναρξη της κρίσης και τις συνέπειες της κρίσης στην Ευρωζώνη. Με χώρες που αντί να συγκλίνουν, να απέκλανουν και περισσότερο, χώρες που έχουν το ίδιο νόμισμα αλλά αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις και μερικά σημεία σύγκλησης, ιδιαίτερα σε θέματα ανταγωνιστικότητας επενδύσεων και χρηματοδότηση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας έλειπαν από το οικοδόμημα. Επίσης κάτι άλλο που είναι απαραίτητο στο, στις σημερινές συνθήκες και δικαίως και εύστοχα υπερβάως είπε ότι άσχετα με την έκβαση του Βρετανικού δημοψηφίσματο, έπρεπε, θα έπρεπε να προβληματιστούμε το θέμα αυτό και όχι μόνο να προβληματιστούμε, αλλά να δώσουμε και μια απάντηση. Πολλό δε μάλλον που το δημοψήφισμα είχε τη γνωστή, το γνωστό αποτέλεσμα και θα πρέπει η Ευρωζώνη να δώσει μια εικόνα ισχύω, πρωτοβουλία και ικανότητα και δυνατό, να αντιμετωπίσει τι σημερινέ προκλήσει. Γι' αυτό και χρειάζεται προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Περί αυτού δεν έχω κανέναν ενδιασμό. Το πιστεύω ακράδαντα και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που έχει αυτή τη γνώμη. Και μάλιστα προσπαθήσαμε με τον ένα ή άλλο τρόπο να θεσπίσουμε τέτοιου είδους προϋπολογισμό. Τέτοιου είδους λέω, γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, είναι μία μορφή ε, ε συγκέντρωσης κάποιων δημοσιονομικών μέσων προκειμένου να εξασφαλιστεί απαραίτητη αλληλεγγύη υπό όρους. Και βλέπουμε ότι ο λόγω μηχανισμός ακόμη και αν ε, υπόκειται συγκεκριμένη διαχείριση, θα μπορούσε να είναι ένα ε, προκαταρκτικό σχέδιο, ίσως ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου ή ενός ε, Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού της Ευρωζώνης, με τη στήριξη βέβαια κάποιων απαραίτητων μηχανισμών. Και στις, στη Δημοσιονομική Βούληση που εκδηλώθηκε, για παράδειγμα, στις επενδύσεις του επενδυτικού σχεδίου Juncker, και αυτές αποτελούν την έκφαση της απαραίτητης ικανότητας δημοσιονομικής δράσης και μάλιστα ισχυρής δημοσιονομικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστούν κάποιες οικονομικές καταστάσεις που ίσως έχουν αντικυκλικό χαρακτήρα ή μπορεί να ε, διευρύνουν ένα κύκλο που έχει προβλήματα στην αναζωογόνησή του. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που μας προβληματίζουν και που δεν έχουμε ήδη από τώρα όλες τις απαντήσεις, αλλά σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε μη τι άλλο τις ερωτήσεις. Και μια και χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε και ένα μέσο, όχι μόνο να τον καταρτήσουμε, αλλά και να τον ελέγξουμε. Και αν υπάρχει προϋπολογισμό, σημαίνει ότι θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να συζητήσει αυτόν τον προπολογισμό, να τον εγκρίνει, γιατί δεν βλέπουμε ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιο προπολογισμό χωρί τον απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο. Γιατί αυτό ο δημοκρατικό έλεγχο μπορεί για, για πολλούς πολίτες των χωρών μας φαίνεται μακριά, απο, απομακρυσμένος από την πραγματικότητα, χωρί όμω κανένα τέτοιο δημοκρατικό έλεγχο θα ήταν πολύ προβληματικό κάτι τέτοιο. Τώρα, και αν έχουμε ένα προπολογισμό, χρειαζόμαστε και κάποιον που θα έχει τη δυνατότητα να τον εκτελέσει κιόλα, να τον εφαρμόσει. Και είναι γνωστή και η συζήτηση η σχετική. Ε, παρά τους ενδιασμούς ε, που υπάρχουν. Γιατί ε, μερικοί μιλούν για διαχείριση σε αμυγός κοινοτική διαδικασία και μέθοδο και άλλοι ε, είναι υπέρ περισσότερο μια διακυβερνητικής μεθόδου και αυτά είναι μείζωνα ζητήματα. Δεν πρόκειται να λάβω θέση γιατί ούτως ή άλλως αυτό το θέμα θα γίνει ιδιαίτερα δύσκολο τους επόμενους μήνες κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν όμως έχουμε προπολογισμό, χρειαζόμαστε και πόρους. Και το θέμα των πόρων είναι απολύτω απαραίτητο. Και μάλιστα οι πόροι αυτοί μπορούν να ισχύουν γενικώ για, τον για τον ενωσιακό προπολογισμό, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερο για τον προπολογισμό μια Ευρωζώνη και θα πρέπει να προσδιορίσουμε το είδο αυτών των πόρων. Και εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε διάφορε λύσει. Ίδιου πόρου, ένα τμήμα που θα προέρχονται από τους εθνικούς. Πάντως τέτοιους πόρους χρειαζόμαστε για να καταρτήσουμε τέτοιο προϋπολογισμό. Και θα ολοκληρώσω εδώ με μία πεποίθηση, γιατί θέλω να αφήσω και τους άλλους συναδέλφους να μιλήσουν. Ε, ξεκινούμε αυτή τη συζήτηση με θεσμικό τρόπο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Μόνο με το θεσμική μέθοδο δεν θα βρούμε το σωστή διέξοδο. Αν ε, επισέλθουμε στη συζήτηση πολιτουργική σκοπιά, συγκεκριμένη, σαφή, πού είναι τα προβλήματα, ε, τι, προβλήματα θα μπορούσε να επιλύσει ένας τέτοιος προϋπολογισμός, τι δυνατότητα δράση μας δίνει, ταχείας δράσης, γιατί οι λαοί μας χρειάζονται απτές λύσεις και εξασφάλιση ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα της Ευρώπης με συγκεκριμένες πολιτικές. Και αντί να επισέλθουμε από την θύρα τη θεσμική, που ίσως θα χρειαστεί κάποια στιγμή γιατί όλα θα έχουν τέτοια απεικόνηση και θεσμική και θα επηρεάσουν τη θεσμική λειτουργία, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να, περάσουμε και από την ε, πιο χειροπιαστή θύρα, τη θύρα την επιχειρησιακή, τη λειτουργική, τι επενδύσεις θα χρειαστούν, τι εξασφαλίσεις ε, η ασφάλεια ανεργίας ή τι είδου ευρωπαϊκή ικανότητα να εξασφαλίσει ένα στρώμα αλληλεγγύης για θέματα ενεργείας, για παράδειγμα. Μόνο με τέτοια χειροπιαστά θέματα και προτάσεις θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα των διακυβευμάτων στους ε, πολίτες μας. Αλλιώς θα χαθούμε σε αυτό το λαβύρινθο της ε, θεσμικής συζήτησης ε, που μας απομακρύνει από τον προβληματισμό και τις ανησυχίες των πολιτών μας που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να μας δείξουν την εμπιστοσύνη τους. Thank you. Σας ευχαριστώ και Τσακαλώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ρομπέρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επιτροπή του Κοινοβουλίου και τη δουλειά που κάνει πάνω στο θέμα. Είναι ένα θέμα κρίσιμο και θα ήθελα να αναφέρω τρεις λόγους για τους οποίους πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης. Πρώτον, ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Ορισμένες φορές έχω ασκήσει κριτική στις ε, προβλέψεις ανάπτυξης της Κομισιόν και της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όταν έχουν δηλώσει του στυλ η ανάπτυξη δεν πάει πάρα πολύ καλά γιατί η παγκόσμια οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά και μπορεί να τα πάμε χειρότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Βολιβία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι μια μικρή κλειστή ε, ανοιχτή οικονομία, είναι μια μεγάλη οικονομία. Οπότε αν η παγκόσμια οικονομία δεν τα πάει καλά, ίσως ένας λόγος είναι ότι η Ευρώπη δεν κάνει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε, είχαμε στο παρελθόν διάφορες περιοχές του κόσμου που δεν τα πήγαιναν τόσο καλά. Και στο μέλλον μπορεί η Ασία να τα πάει καλύτερα ή χειρότερα, η Αμερική το ίδιο. Όταν κάποια περιοχή τα πάει χειρότερα πρέπει μια άλλη περιοχή να γεμίσει το κενό. Αν είναι λοιπόν η Ευρώπη να παίξει τον ρόλο της, δεν μπορεί απλά να έχει πλεονάσματα τρευσών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά έχει μια ευθύνη για την παγκόσμια ζήτηση με έναν τρόπο που δεν έχει μια μικρή ανοιχτή οικονομία. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον αυτόματο ρόλο ε, ενό προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Εάν παραδείγματο χάρη υπάρχει ύφεση στο Τέξα, ε, πηγαίνουν οι πόροι του Ομοσπονδιακού Προπολογισμού στο Τέξας. Ε, δηλαδή πληρώνει το Τέξας λιγότερους φόρους και υπάρχουν και επιδοτήσεις. Αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Εάν ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός χρηματοδοτεί αυτούς τους αυξημένους πόρους μέσω δανεισμού και έκδοσης ομολόγων, οι Τεξανοί αποζημιώνονται από το σύνολο των Αμερικανών. Τα ομόλογα αυτά αποπληρώνονται είτε είναι κανείς από την ε, Μασαχουσέτη, την Καλιφόρνια κτλ. Οπότε υπάρχουν δύο αποτέλεσματα. Αυτό το οποίο λένε σταθεροποιητικό οικονομολόγοι, δηλαδή μια χώρα έχει ένα σοκ ασύμετρο και πέφτει σε ύφεση και το άλλο είναι ότι υπάρχει το φαινόμενο αυτό της ε, εξίσωσης, δηλαδή ενός είδους ε, αλληλεγγύη. Σήμερα θα είναι σε ύφεση το Τέξας, αύριο θα είναι η Μασαχουσέτη και θέλουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη όπου θα Σημαίνει το ίδιο, ότι μία στιγμή θα έχει Ελλάδα κρίση, την επόμενη Γερμανία, την άλλη θα είναι η Φιλανδία ή η Πορτογαλία. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι για να ασκείται δημοσιονομική πολιτική. Σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια που θα υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε το κατάλληλο πόσο ζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα εξωτερικά μεγέθη. Το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι η Γαλλία θα ήθελε παραδείγματο χάρη να επεκταθεί, αλλά η επέκταση αυτή θα ωφελήσει την Γερμανία και την Πορτογαλία. Και ή μπορεί να ήθελε να κάνει η Πορτογαλία και η Γερμανία το ίδιο, αλλά τα ωφέλη όσον αφορά ε, θα είναι εισαγωγές από άλλες χώρες. Οπότε η λύση είναι να επεκταθούν όλες οι χώρες μαζί. Οι εξωτερικότητες να εσωτερικοποιηθούν. Και είναι σαφές, για μένα τουλάχιστον, πως ε, υπάρχει μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, την οποία θα χρειαζόμασταν με τα επίπεδα αυτά τα υψηλά της ανεργίας, η οποία όμως δεν λαμβάνει χώρα γιατί δεν υπάρχει χώρος, όπως είπαμε, να ιστορικοποιηθούν οι εξωτερικότητες. Αν δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, τι έχουμε. Αν δεν είμαστε νομισματική ένωση με την έννοια που είναι η Γερμανία, ο Καναδάς, η Γερμανία σε σχέση με τα Λέντερ, όπως είναι η Αυστραλία. Τι έχουμε, έχουμε νομισματική πολιτική που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σύμμετρα σοκ, τους ε, κραδασμούς, ούτε καν και συμμετρικά δεν νομίζω να μπορεί να αντιμετωπίσει αν δεν δούμε το ζήτημα του χρέους γιατί ε, πλέον δεν λειτουργεί σχεδόν η νομισματική πολιτική. Δηλαδή μπορεί να μειώνει τα επιτόκια τη η Κεντρική Τράπεζα αλλά αυτό δεν επηρεάζει την Ισπανία ή την Πορτογαλία ή την Ελλάδα. Αλλά υποθέσουμε ότι έχουμε νομισματική πολιτική, δεν έχουμε πολιτική υποτίμηση και δεν έχουμε δημοσιονομική πολιτική αν δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Τι υπάρχει λοιπόν, το ύψο του μισθού. Είναι ο μόνος τρόπος να απορροφηθούν κραδασμοί στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά σε σχέση με τον ευρωσκεπτικισμό. Μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει όταν ο μόνος τρόπος να απορροφηθούν τα σοκ είναι η μισθή. Και η Μισελ εδώ πέρα έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Μια νομισματική ένωση που δεν θα βασίζεται μόνο στο να απορροφούν οι μισθοί τους κρατασμούς, αλλά και μια νομισματική ένωση η οποία θα έχει τα οικονομικά εργαλεία τα οποία θα παίζουν το ρόλο της ε, υποτίμησης, όπως η δημοσιονομική πολιτική, υπό δημοκρατικό έλεγχο. Αν θέλουμε όντως να καταπολεμήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό τα χρόνια ε, μετά από το Brexit, αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι θα αισθάνονται ότι δεν είναι μόνο οι μισθοί αυτοί οι οποίοι θα απορροφούν τους κραδασμούς και ότι δεν θα είναι μόνο ελαστικοί προς τα κάτω αλλά και προς τα πάνω και θα πρέπει η πολιτική αυτή να είναι ή υποδημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία. Νομίζω πως αυτός είναι ο τρόπος να αποφύγουμε τον ευρωσκεπτικισμό. Και εμείς που είμαστε υπέρ της Ευρώπης χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πυγμή που θα λέει ναι έχουμε πανευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτό θα βλέπει ο κόσμος και πράγματι λειτουργούν και είναι, δίνουν δοσία δημοκρατικά. Σας ευχαριστώ κύριο Σπαντών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ την έκθεση που συντάξατε και, έχει, και γιατί έχει μια ευρύτερη προσέγγιση από αυτή του τίτλου της. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή να μιλήσουμε για την διακυβέρνηση και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της Ευρωζώνης που πρέπει να ενισχύσουμε και λόγω των ε, γεγονότων που έχουν ε, αυξήσει το, την αβεβαιότητα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Ε, έχω πολλά κοινά λοιπόν με την έκθεση. Θα ήθελα να μπω σε κάποιες από τις αρχές εντάχει που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες για να δούμε πώς θα βελτιώσει την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνη. Καταρχάς, προφανώς, όταν μιλάμε για τις πολιτικές Ευρωζώνης θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο, στις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικές φορές δίνει την εντύπωση ότι παρότι είμαστε μέλη μιας ένωσης ε, και ενός ε, σφιχτού συστήματος, ο μόνος μηχανισμός ε, προσαρμογής, και αναφέρθηκε ο Ευκλήδης αυτό, είναι το εθνικό επίπεδο, οι εθνικοί μηχανισμοί. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη ευρωπαϊκών εργαλείων πέρα από τις επιλογές της πολιτικής. Και μπορώ να σκεφτώ διάφορες περιπτώσεις όπου αυτό αποδεικνύεται αληθινό. Δεύτερον, το οποίο απορρέει από το πρώτο, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στην Νομισματική Ένωση, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε δύο τροχίες, ε, παράλληλα και αμφίδρομα. Ο επιμερισμός των κινδύνων και ο μετριασμός των κινδύνων. Το ακούσατε όταν συζητήσαμε για την ε, Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι είναι μια γενική αρχή, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς. πίν και στην απασχόληση και στις πολιτικές για την αγορά εργασίας. Και θα προσπαθήσω να σας το ξεκαθαρίσω σε λίγο αυτό. Τρίτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τα κίνητρα μέσω της πολιτικής με βάση αυτές τις δύο ε, προναφερθήσεις αρχές. Εγώ, Φερρυπίν, είμαι υπέρ των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπίσουμε ε, την μακρο, μακρόχρονη χαμηλή ανάπτυξη. Φυσικά, οι μεταρρυθμίσεις είναι τμήμα της λύσης. Το θέμα όμως ε, που πρέπει να μας απασχολήσει ως πολιτικούς είναι ποια είναι τα κίνητρα που έχουν οι πολιτικοί για να εισαγάγουν τι διαρθωτικές μεταρρυθμίσει. Και εδώ, σχεδιάζοντας τα εργαλεία της πολιτικής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο. Λέω πάντα ότι το θέμα της ε, ευελιξίας δεν είναι το πώς ε, μια κυβέρνηση θα ακολουθεί όλο και λιγότερο τους κανόνες. Αντίθετα, πώς θα δίνουμε περισσότερα κίνητρα είναι το θέμα για να υπάρξουν ε, διευθυντικές μεταρρυθμίσεις από τη διαφθορτική πλευρά ή από τη μακροπρόθεσμη ζήτηση, αυτό είναι το ένα τμήμα. Χρειάζεται και μακροπρόθεσμη ζήτηση. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία σε μακροοικονομικό επίπεδο. Θα ήθελα ιδανικά να έχω μία ευρωπαϊκή μακροοικονομική πολιτική και μία δημοσιονομική ικανότητα που να στρέφεται και να κεντράρει στην ζήτηση και πώς θα μπορούσαμε να αναδιανύμουμε την δημοσιονομική ικανότητα στις χώρες Ευρωζώνης. Αν γίνει σωστά αυτό, τότε η, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μακροοικονομικές πολιτικές και στις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο πράγματα, επαναλαμβάνοντας μια πρόταση που έχει κάνει η Ιταλική κυβέρνηση, η οποία δεν είναι καινούρια. Είναι ένα κλασικό οικονομικό εργαλείο. Είναι η εισαγωγή ενός ε, συστήματος ε, ε, επιδομάτων ενεργείας στην Νοησματική Ένωση. Γιατί? Ένας από τους λόγους που ανέφερε ο Ευκλήδης είναι ότι αν έχεις μια νομισματική ένωση, τότε δεν υπάρχει σωστή, σωστό εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής για να απορροφήσεις τα σοκ. Επομένως, τι σημαίνει η αγορά εργασίας. Φυσικά μπορεί να υπάρξει προσαρμογή στους μισθούς ή στα επίπεδα ανεργίας. Και φυσικά και τα δύο είναι, συνδέονται μεταξύ τους. Εάν θέλεις να έχεις ε, μια φιλική ε, προς την απασχόληση και στην απορρόφηση νομισματική ένωση, θα πρέπει να έχεις μηχανισμούς απορρόφησης όταν έχεις ασύμετρα σοκ. Ένας άλλος λόγος που πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τους κανόνες της πολιτικής σε μια νομισματική ένωση και σχετίζεται με την ανεργία, είναι ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κυκλική ανεργία, ούτως ώστε να αποφύγουμε ότι η κυκλική ανεργία τελικά παραμένει α, για μεγάλο χρονικό διάστημα και γίνεται διαρθωτική και ε, προκαλεί λιγότερη και όχι περισσότερη σύγκληση. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι γιατί έχει νόημα να κάνουμε μια συζήτηση ε, για το πώς θα ξανασχεδιάσουμε την νομισματική ένωση, ούτως ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά εργασίας και στο θέμα της απασχόλησης. Ειδικά επειδή συνδέονται με το πώς ε, λειτουργούν ε, οι μακροοικονομικές πολιτικές στην Νομισματική Ένωση. Κάτι άλλο, ε, το οποίο μου άρεσε στην έκθεση. Αν έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να αντιμετωπίζει σωστά τα, τους ασύμμετρους κραδασμούς. Αλλά μην ξεχνάμε και τους συμμετρικούς κραδασμούς, δηλαδή αυτούς που πλήττουν όλη την νομισματική ένωση. Και νομίζω εδώ ότι οι προτάσεις που κάνανε για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, κινητοποιώντας τους ε, υφιστάμενους πόρους, παραδείγματο χάρη ε, μέσω του μηχανισμού σταθερότητας, είναι σημαντικό. Οι επενδύσεις επίσης είναι ένα συνδυασμό πολλών παραγόντων. Υπάρχουν επενδύσεις, αν υπάρχει αίσθηση ότι περιμένεις η ζήτηση να αυξηθεί στο μέλλον ε, και μάστα με κέρδος, γίνονται επενδύσεις εάν η τα εμπόδια σε επενδύσεις που οφείλονται στα διαφορετικά προβλήματα αρθούν. Και υπάρχουν επενδύσεις αν έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον, το οποίο συμπεριλαμβάνει και εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα που θα υπάρχει στο μέλλον και στους θεσμούς που θα υπάρχουν. Κάτι νομίζω που ξεχνάμε και μας λείπει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Pierre Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με συγχαρητήρια προς τους ε, διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας ε, και την ευχαρίστησή μου και την... ευχαριστήρια για την πρόσκληση. Είχαμε και πέρυσι συναντηθεί με πολλούς ευρωβουλευτές κατά την κατάρτιση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και μάλιστα όλα έγιναν σε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η, ιστορία, η ευρωπαϊκή ιστορία ε, είναι, γίνεται σταδιακά και όπω είπε και ο Μισελ Σαπά, έχουμε μια οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά φαίνεται δημιουργήσαμε ένα προθύστερο σχήμα, ε, δηλαδή αποφασίσαμε πολιτικά ότι θέλουμε ένα κοινό νόμισμα και προσπαθήσαμε να το κάνουμε χωρίς να έχουμε ουσιαστικά κοινέ οικονομικές πολιτικές. Δηλαδή, μας πρόλαβε βέβαια η ιστορία, η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση και αναγκαστήκαμε να προσπαθήσουμε να χάσουμε το, να κερδίσουμε το χαμένο έδαφο, συγγνώμη, και αυτό κάναμε τον τελευταίο καιρό με την ενίσχυση της, των πολιτικών σταθερότητα και ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή μας οικοδόμηση στον οικονομικό και νομισματικό τομέα είναι ένα πραγματικό ψηφιδωτό, από το οποίο λοιπόν πολλές ψηφίδες. Και από εμά αναμένεται, σε εμά εναπόκειται να τη συμπληρώσουμε. Και αρκεί να λάβουμε το παράδειγμα του Ρομπέρ Σουμάν που έλεγε ότι το δημιουργ... η ευρωπαϊκή οικοδόμηση δεν θα γίνει εν μία δεν θα γίνει μόνο μιας, με μια μονοκοντιλιά. Και ακριβώς ε, στη θέση του ερωτήματος ε, για το αν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό προπολογισμό με ίδιους πόρους, ε, φυσικά αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, ένας μακρόπνοος στόχος. Και αν λάβουμε αυτό το σημείο, σημείο φετηρίας του συλλογισμού, ίσως κάπου χαθούμε στην πορεία. Οπότε η δική μου πρόταση θα ήταν να επιλέξουμε θέματα εφικτής αλληλεγγύης, πιθανής αλληλεγγύης και προοδευτικά σταδιακά να οικοδομήσουμε αυτή την αλληλεγγύη. Και φυσικά θα πρέπει να υποτιμούμε την δινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Όχι μόνο εξαιτία ή ε, λόγω του ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος, του βρετανικού δημοψηφίσματος, αλλά γενικώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε 28 χώρε σήμερα, 27 χώρε αύριο ε, για να συμφωνήσουμε μια κοινή φορολογία. Ερωτηματικό. Μία ε, ερώτηση, ένα θέμα είναι ότι η Ευρωζώνη με 19 μέλη έχει ήδη περισσότερη αλληλεγγύη. Το θέμα είναι πώς, ε, ποιο είναι το σωστό πρίσμα, ποιο είναι η σωστή σκοπιά και πώς θα το καταφέρουμε. Καταρχήν, ε, προσπαθώντας να ελεγχιστοποιήσουμε τους φόβους ε, και τις ανησυχίες των μεν και των δε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που αναφέρθηκε. Είναι η μετατροπή αυτής της αξιέπαινης αλληλεγγύης σε μια ευρωπαϊκή ζώνη μεταφορών, μεταφορών κονδυλίων. Είναι σαφές ότι οι χώρες ε, που τα πάνε καλά, οι χώρες που σέβονται όλους τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, είναι σίγουρα έτοιμε να επιδείξουν κάποιο βαθμό αλληλεγγύη, υπό τον όρο όμω ότι χώρε που δεν τα πάνε τόσο καλά ή που βρίσκονται σε κάπω δύσκολη θέση στα θέματα του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και αυτέ θα καταβάλουν τι απαραίτητε προσπάθειε. Μεταξύ αυτών των δύο πόλων θα πρέπει να βρούμε κάποια κοινά σημεία. Εξού και αυτό που μας είπε ο κύριος Παντοάν, ένα σημαντικό θέμα, να έχουμε παράλληλες τροχές ε, όπου θα έχουμε αφενό τη μείωση των κινδύνων που θα συνοδεύεται όμως από έναν επιμερισμό των κινδύνων. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο σταδιακά, προοδευτικά, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο. Είναι σαφές ότι όλοι φέρουμε και εθνικές ευθύνες για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε και παράλληλα εφόσον ε, εξασφαλιστεί μεγαλύτερο σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητα Ανάπτυξη και από περισσότερε χώρε, θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε περισσότερο, να προχωρήσουμε περισσότερο και στο θέμα τη ελληνική. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται και στο εξαιρετικό έγγραφο. Το ταμείο αυτό για τι δύσκολε μέρε, για τα πρόβλεπτα γεγονότα, το Rainy Day Fund σε περίπτωση συγκυριακών κραδασμών, ακόμη και σε περίπτωση όμως αντικυκλικών κραδασμών, μπορώ να φανταστώ ένα, μια τέτοια ελεγγύη που θα έχει προσωρινή βάση. Δηλαδή θα έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση απρόβλεπτη που θα χρήζει ε, προσωρινή ενίσχυση. Αλλά να καταστήσουμε κάτι τέτοιο οριστικό και μόνιμο θα είναι κάπως πιο δύσκολο. Αυτά και βάζω εδώ τελεία για να αφήσουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Um... σε ευχαριστώ ο Έντουαρτ Σικλούνα. Thank ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Όταν ήμουν ε, Ευρωβουλευτής, με ρώτησαν τι έκανα πριν και έλεγα στο πανεπιστήμιο και μου λέγανε «Α, καταλάβαμε». Στη θεωρία ζούσατε εδώ, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών μου λένε τι έκανα πριν, ε, τους λέω ήμουν ε, και μου λένε το ίδιο. Α, εκεί πέρα ε, είχατε ιδέες και διάφορα τέτοια, εδώ είμαστε πιο πρακτικοί και αντιμετωπίζουμε τα άμεσα προβλήματα. Οπότε είναι ενδιαφέρον να διαβάζω αυτή την έκθεση της συναδέλφου της Περβάος και του κυρίου Μπέγκε. Και βλέπω ακριβώς τις ε, διαφορετικές οπτικές. Είναι θέμα οπτικής πράγματι. Συμφωνούμε στο τι θέλουμε να κάνουμε σαν ένα καλό γάμο. Το ιδεώδες θα είναι η τέλεια αγάπη και το να μην είμαστε εγωιστές. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Αλλά ξέρετε οι γρήγοροι και γάμοι υποπίεση συχνά καταλήγουν σε διαζύγιο. Λοιπόν, τα θεσμικά όργανα τα οποία έχουμε σήμερα, το Σύμφωνο Σταθερότητας, η Συνθήκη για τη Σταθερότητα και τον Συντονισμό, το Ευρωπαϊκό Εξάμνο, όλοι αυτοί είναι μηχανισμοί που ασχολούνται με ζητήματα βιωσιμότητας και συντονισμού της πολιτικής. Όμως, πρέπει να τα αφήσουμε αυτά να λειτουργήσουν να οριμάσουν, να εφαρμοστούν πριν να αρχίσουμε να εφευρίσκουμε συνεχώς νέα θεσμικά όργανα. Ο Brexit δείχνει ξεκάθαρα πως ε, δεν είναι δεδομένη η Ένωση. Δεν έχει ούτε μία σχέση με τις ε, ΗΠΑ. Και η απάντηση είναι να, αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε και άλλα θεσμικά όργανα για να πάμε σε πλήρη ενοποίηση. Αλλά και πάλι το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί ε, η ηρωνία είναι ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει δει τα αποτελέσματα του τωρινού, του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Ας δούμε το διπλό και το εξαπλό σύμφωνο. Θα θυμάστε, όταν τα συντάσαμε αυτά εδώ πέρα έχει καταγραφεί η άποψή μου στα πρακτικά που έλεγα ότι αυτά τα πρόστιμα ήταν δρακόντια. Γιατί θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως και σε χώρες οι οποίες θα έχουν ήδη πρόβλημα. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και μετά τους ρίχνουμε και πρόστιμο πάνω. Και η απάντηση ήταν ναι, μα δεν θέμε να επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν με τη Γαλλία και τη Γερμανία που παρέβηναν τους κανόνες και δεν έτρεχε τίποτα. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και αυτή τη φορά θα είναι τόσο σοβαρά τα αποτρεπτικά μέσα που καμία χώρα δεν θα τολμήσει να φτάσει εκεί. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει σε, στο σημείο δύο χώρες ε, να λέει η Κομισιόν ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες, οι χώρες δεν το δέχονται. Αλλά το συζητήσαμε στο Συμβούλιο και αύριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Το θέμα της ευελιξίας, ε, του κενού αυτού της ε, παραγωγής, ε, της παραγωγικότητας, αν το μετράμε σωστά. Όλοι ε, προτείνουν νέους δείκτες για να αντικαταστήσουν τους κανόνες για το έλλειμμα, πως θα πρέπει να είναι κάποιος κανόνας για τις δαπάνες. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και δεν έχουμε δει ακόμα την σωστή εφαρμογή των υφισταμένων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και με τα όσα συμβαίνουν με την Τραπεζική Ένωση που μιλάμε για Μπέιλιν και γιατί λέμε δεν θα ξαναγίνει ποτέ διάσωση και κανένα κράτος δεν θα πρέπει να ξανασώσει τράπεζα. ρωτήστε και τον συνάδελφό μου, τον Πιερ Κάρλο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή το μία λύση για όλους δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τυφλό σύστημα το οποίο θα λειτουργεί αυτομάτως. Μπορούμε να Έτσι θα δημιουργήσουμε χειρότερες κρίσεις από αυτές που προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Οπότε η πρότασή μου είναι ας αφήσουμε λίγο να εργαστούν τα θεσμικά όργανα και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τα καλά τους και τα κακά τους. Όταν ακούω δηλαδή για σύγκληση και εφαρμογή, ε, σε σύγκληση σε φορολογία, κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ε, έτσι μπορεί μια χώρα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και εμείς με τον ενθουσιασμό μας. Ε, ναι, εντάξει, συμφωνούμε όλοι ότι μια μέρα αυτός είναι ο στόχος, αλλά δεν μπορούμε να βιαζόμαστε. Και οι λαοί μας δεν έχουν δει ακόμα τι έχουμε οικοδομήσει, δεν το έχουν δει να λειτουργεί και να έχει αποτελέσματα για να προχωρήσουμε με τρόπο φυσικό στο επόμενο βήμα. Οπότε, ε, εγώ δεν ε, εκφράζω μια ευρωσκεπτικιστική άποψη. Θα συμφωνούσα πως ε, η Ένωση θα γίνει πλήρης, θα υπάρξει ένα Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Αλλά ας δούμε πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία έχουμε ήδη δημιουργήσει, ας τα αφήσουμε να λειτουργήσουν και μετά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, Γερούν. Ο Γερούν Τάισελγκλουμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε εδώ την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ τα δύο μέλη τους δύο προβουλευτές δηλαδή που ετοίμασαν αυτή την έκθεση. Τους μίλησα πριν από κάποιες εβδομάδες ή κάνα μήνα ίσως. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κανενα μηνα ισως νομιζω οτι ειναι παρα πολυ σημαντικη η δουλεια σας. Βασίστηκε στην έκθεση των πέντε προέδρων και στα όσα εμπεριέχει αυτή. Φυσικά, πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν. Στην έκθεση των πέντε Προέδρων είπαμε ότι στο τέλος του 2016 θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να δώσει συνέχεια στην έκθεση και να κάνει την πιο τεχνική και αναλυτική δουλειά για να οικοδομήσουμε τα εργαλεία για τη δεύτερη φάση της έκθεσης. Εσείς ξεκινήσατε με τη δική σας έκθεση που εξετάζουμε σήμερα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη. Η δημοσιονομική ικανότητα είναι κάτι που θέλουν πολύ στη δημόσια και πολιτική συζήτηση μία ΟΝΕ, ναι. καλό είναι να την έχει. Αλλά για πολύ διαφορετικούς λόγους πιστεύουν οι μεν από τους δε. Ορισμένους από τους λόγους αναφέρονται και στην έκθεσή σας. Από τον Τίμπεργ, τον Ολλανδό ε, οικονομολόγο, ε, ο οποίο έχει πάρει και βραβείο Νόμπελ, είναι ότι αν έχει πολλά εργαλεία, μερικέ φορέ μπορεί να δυσκολεύεσαι, να δυσκολευτεί. σω γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πιο πολύ, μήπω ε, περιμένουμε πάρα πολλά, έχουμε πολλέ προσδοκίε από ένα και μόνο εργαλείο. Θα υπάρξει ανταγωνισμό ε, για την ε, χρήση των διαφόρων εργαλείων. και αν θέλουμε να υλοποιήσουμε πολλού στόχου σε πολλού τομεί, πρέπει να διαλέξουμε τα εργαλεία μα. Επίση, σε τι θα πρέπει να τον ξοδεύουμε τον προπολογισμό. Η έκθεση μιλάει για τρεις βασικούς τομείς. Καταρχάς είναι να δώσουμε κίνητρα για διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, αναφέρεται εκτενώς και στην έκθεση των πέντε προέδρων. Αλλά νομίζω η σειρά είναι αντίστροφη. Λέμε ότι περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει σε διορθωτικό επίπεδο για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής σύγκλησης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και μετά από αυτή τη σύγκληση, που είναι ουσιαστικά αντιστροφή των αποκλήσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια, μετά από αυτή τη σύγκληση μπορούμε να πάμε στα επόμενα βήματα ε, για να υπάρξει σύγκληση των πολιτικών. Για να ολοκληρώσουμε την ε, νομισματική ένωση. Εδώ, αν κατάλαβα καλά, η έκθεση λέει κάτι που με εντυπωσίασε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ότι αν θέλετε σύγκληση, χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία για να δρομολογήσουμε τη διαδικασία σύγκληση. Αν δω που είμαστε τώρα, οικονομικά και πολιτικά, είναι μια προσέγγιση εντυπωσιακή. Μια πιθανή επίσης λειτουργία το μέσο αυτού θα ήταν να αντιμετωπίσει τους ασύμμετρους κραδασμούς. Νομίζω ότι στην Ευρωζώνη υπήρξαν πολύ λίγοι ε, ασύμμετροι κραδασμοί. Οι κύκλοι της οικονομικής δραστηριότητας ήταν εντυπωσιακά συμμετρικοί. Ε, εκεί που έχουμε συμμετρία είναι σε επίπεδο εθνικών πολιτικών. Η χρηματοπιστωτική κύκλη από την άλλη είναι πολύ πιο αποκλίνοντες. Και με αυτό δεδομένο ο Καλύτερο τρόπος για να ε, ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα απορρόφηση των κραδασμών είναι να ολοκληρώσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαιογορών. Το έχω ξαναπεί αυτό και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ότι για να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα απορρόφηση των κραδασμών στην Ευρωζώνη, οι οικονομίε τη Ευρωζώνη χρειάζονται μηχανισμού που θα επιτρέπουν στον ιδιωτικό τομέα να παίξει το ρόλο του της απορρόφησης των κραδασμών. Γι' αυτό η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση των Κεφαλαγορών ε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Επίσης, ο κίνδυνος των συμμετρικών σοκ σημαίνει ότι θα πρέπει οι εθνικοί μας προπολογισμοί να έχουν ένα περιθώριο, ένα αποθεματικό. Βγαίνοντα βέβαια σε μια κρίση όπω αυτή που γνωρίσαμε, είναι πολύ εύκολο να το λε, αλλά δύσκολο να το κάνει. Και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε εθνικό επίπεδο ε, που οι προπολογισμοί είναι πολύ ψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, έχουμε αυτό το περιθώριο, αυτό το αποθεματικό. Αυτό είναι ο μακροπρόθεσμος στόχο για όλους μας. Για την αντιμετώπιση των συμμετρικών σοκ ε, με την δημοσιονομική ικανότητα χρειαζόμαστε περισσότερα, ε, περισσότερους πόρους. Από πού θα έρχονται όμως είναι το ερώτημα. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ε, που είναι ένας ε, μηχανισμός δανειοδότησης. Δεν έχει δικά του μέσα. Δεν, έχει, δεν συγκεντρώνει φόρους. Δεν λέει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις έτσι το θέμα του από πού προέρχονται τα χρήματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα θέματα. Το τι κάνουν τα εργαλεία λοιπόν, πώς τα χρηματοδοτούμε. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν και νομίζω ότι σήμερα είναι καλή ευκαιρία για να τα συζητήσουμε. Έπειτα υπάρχει και η πολιτική διάσταση. Πιστεύω ότι σήμερα το πρωί έγινε μια συζήτηση, μια διάσκεψη της Σλοβακικής Προεδρίας για την ανεργία και για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης της ανεργίας. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα σα. Στη χώρα μου τουλάχιστον το σύστημα κοινωνική ασφάλισης και το συνταξιωτικό σύστημα ιστορικά και πολιτιστικά μέσα από τη δουλειά που έχουν κάνει γενιές έχουν φτάσει στη σημερινή μορφή. Ε, οι κοινωνικοί εταίροι ε, είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν σήμερα τα επιδόματα ανεργία στη χώρα μου. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται και με την κουλτούρα και με την παράδοση. Ε, το αν ένα πράγμα, ένα πράγμα μπορεί ας πούμε, οικονομικά να είναι ενδιαφέρον ω ιδέα. Το θέμα είναι οι χώρε τι μπορούν να κάνουν. Και στο σημερινό, στη σημερινή συγκυρία, στο σημερινό πλαίσιο, είναι μια πρόκληση. Στην ε, Ολλανδία ένα θέμα που μας απασχολεί είναι ότι αν ε, η Ευρώπη αρχίσει να μπερδεύεται στα ασυντιοδοξιδοτικά μας, θα εξαγριωθούν οι Ολλανδοί, γιατί είναι ε, ένα τμήμα τη ταυτότητα ε, του κοινωνικού μας συστήματος. Ε, είναι τεράστιο βήμα αυτό. Για να περάσουμε σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπισης Ανεργίας, αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ σταδιακά. Είναι ενδιαφέρον ιδέα για το μέλλον, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη οικονομική και θεσμική σύγκληση πριν φτάσουμε εκεί. Ας συνεχίσουμε τη δουλειά, ας συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ας αρχίσουμε την οικονομική σύγκληση. Κάποτε η Ευρώπη ήταν μια μηχανή σύγκλησης. Ας, δούμε, ας δούμε και ας προωθήσουμε αυτή τη σύγκληση πριν πάρουμε τα επόμενα βήματα για μεγαλύτερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση. Ο Πέτρ Καζιμίρ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση και να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο για την πρόσκληση ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι είμαι εδώ ω υπουργό Οικονομικών και όχι ως εκπροσωπών την Προεδρία του Συμβουλίου, ω Πρεζιντέντε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη πρέπει να αρχίσουν ειλικρινεί συζητήσει για το μέλλον. Και το θέμα των μακροοικονομικών σταθεροποιητών είναι ε, τμήμα αυτή τη συζήτηση, αναπόφευκτο, αναπότραστο τμήμα και τη μελλοντική συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι για τα θέματα αυτά χρειαζόμαστε συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Και νομίζω ότι είναι αναφίβολο ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη αυτή η συζήτηση. Δεν είμαι αφελής, δεν περιμένω ρηξικέλευθη πρόοδο τους επόμενους μήνες, αλλά είμαι έτοιμος ε, να εξετάσουμε ε, ανα πάσα στιγμή κάποιες προτάσεις και λύσεις. Και διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη η δημοσιονομική ικανότητα είναι ένα ζήτημα μέσοπρόθεσμο. Αλλά αυτό που σήμερα αποκαλούμε μεσοπρόθεσμη φιλοδοξία, ίσως ε, μετασχηματιστεί αύριο σε μακρόπνο, μακροπρόθεσμο στόχο. Και από μακροπρόθεσμο θα γίνει του Αγίου Ποτέ ίσως σε λίγα χρόνια να καθόμαστε εδώ στην ίδια τράπεζα, αλλά με πολύ διαφορετική σύνθεση. Αυτό δεν είναι και πολύ βέβαια αισιόδοξο. Υπάρχει σα, σαφής ανάγκη ε, μηχανισμών για την αντιμετώπιση ασύμετρων και συμμετρικών κρατασμών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το θέμα της δημο... δημοσιονομικής ικανότητας είναι ζωτικό στοιχείο μιας σταθερής ευρωζώνης. Και επί τη ευκαιρία για την ευρωζώνη, η σταθερότητα της ευρωζώνης ε, είναι κρίσιμη και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό σχέδιο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, οι δημοσιονομικοί σταθεροποιητέ είναι σημαντικοί άμεσα ή έμεσα για ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Ιδιαίτερα μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό ε, να κρατήσουμε συσπηρωμένες τις υπόλοιπες 27 χώρες μέλη. Και θέλω να τονίσω ότι είναι ε, κρίμα που η πρόταση για κοινούς ε, δημοσιονομικούς μηχανισμούς συνδέονται με την έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχία και την ε, ε, βραδικίνητη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Συμφωνώ επίση ότι η δημοσιονομική ικανότητα μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνο εφόσον η αλληλεγγύη συνδέεται στενά με την υπευθυνότητα. Αλληλεγγύη και ευθύνη. Σαφείς κανόνες θα πρέπει να περιορίζουν τον ηθικό κίνδυνο και τις με... μόνιμες μεταφορές. Επίσης δεν θα πρέπει να χρειάζονται ε, αποφάσεις που θα επαφείται στη διακριτική ευχέρεια. Όπως είπε ο Γιαρούν, ο Γιαρούν ε, είναι αλήθεια ότι συζητήσαμε και αυτό το θέμα των διαφόρων ε, μηχανισμών ή ιδιαίτερα μετά την πρωτοβουλία του Παντοάν στο Μιλάνο και σίγουρα στη διάσκεψη κορυφή την άτυπη τη Μπρατισλάβα θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα ενό ευρωπαϊκού μηχανισμού ή συστήματο για, για την ανεργία. Αλλά είναι σαφέ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα και να δημιουργήσει ένα κεντρικό σύστημα στις Βρυξέλλες, ένα ενιαίο. Εμείς θέλουμε ένα σύστημα που θα είναι συμπληρωματικό στα εθνικά συστήματα και όχι, δεν θα υποκαθιστά ούτε θα αντικαθιστά, αλλά θα προστίθεται στα εθνικά συστήματα αυτό το σύστημα ή ο μηχανισμός ε, για την προστασία από την ανεργία. Και αυτό προς το παρόν είναι βέβαια θεωρητική συζήτηση. Και αυτό είναι ο ρόλος ε, των think tanks. Πολύ ονειρευόμαστε αυτή την καλύτερη και ευφιέστερη ολοκλήρωση στο μέλλον, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι η καιρή είναι πολύ χαλεπή, απαιτητική, για να το πω διπλωματικά, και κατά τη γνώμη μου η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει με ευρία συνένεση για την ανάγκη Μία δημοσιονομική ικανότητα. και την ίδια την ανάγκη τη δημοσιονομική ικανότητα και μετά η συζήτηση για τις ειδικέ λειτουργίες και τα συγκεκριμένα είδη των μέσων, καθώς και το νομικό πλαίσιο. Και αυτό θα ξεκινήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει και με το νομικό πλαίσιο. Αυτά από πλευρά μου και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στις ερωτήσει. των σκιωδών εισηγητών. Πιεζόμαστε χρονικά. Ο καθένα έχει τη διάθεση του δύο λεφτά και θέλω να τα σεβαστεί, παρακαλώ, γιατί αλλιώ θα τα καταφέρουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε στι 9 η ώρα. Ο Σίγκφριντ Μούρισαν από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για μη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, βεβαίως το πρώτο που μου έρχεται είναι γιατί την χρειαζόμαστε και πώς μπορεί να βελτιώσει την ε, κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Και κατά την άποψή μου, για να έχει νόημα μια τέτοια δημοσιονομική ικανότητα, πρέπει να ε, αντιμετωπίσει τις ε, αιτίες της κρίσης, υπερβολικό χρέος, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τις ιδιαιτερότητες που ανέφερε ο κ. Ντάσιμπλουμ. Λοιπόν, για την ανταγωνιστικότητα. Αναρωτιέμαι, πώς θα μπορούσε μια δημοσιονομική ικανότητα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, να οδηγήσει στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται όλα τα κράτη-μέλη που έχουν πολύ καλά περιγραφεί στις ε, συστάσεις αναχώρα. Το ερώτημα προς εσάς λοιπόν είναι ποιες είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται οι χώρες σας όπου θεωρείτε πως ε, κάποια κίνητρα από τη δημοσιονομική ικανότητα θα σας βοηθούσαν. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Σαπέν, γιατί είναι τόσο δύσκολο για την Γαλλία να επιτύχει στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, για τη σύνδεση με το χρέος. Ε, κύριε Πάντοαν, αναφέρατε την ανάγκη περισσότερης ευελιξίας για να εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν βλέπω τη σύνδεση, δηλαδή πολλές μεταρρυθμίσεις δεν κοστίζουν λεφτά και δεν δικαιολογούν άρα υψηλότερο έλλειμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την σύνδεση που κάνετε, γιατί για μένα δεν είναι πρόφανη. Και μια ερώτηση προς όλους τους υπουργούς. Ε, μιλήσαμε για το πού θα ξοδέψουμε τα λεφτά, αλλά δεν ε, είπαμε πού θα τα βρούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι επιλογές χρηματοδότησης βλέπετε για τη δημοσιονομική ικανότητα και ειδικά από τις χώρες οι οποίες είναι καθαροί φορείς. Κύριε Γκραμένια, Ντάισελμπλουμ και ΣΑΠΕΝ, πόσα είναι διατεθειμένα να συνεισφέρουν οι χώρες σας και πώς θα εξηγήσετε στους ανέργους στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία και σε όλα τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πληρώσουν για άνεργους σε άλλες χώρες σε καιρό κρίσης. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Ντάσιμπλουμ, οι περισσότερες από τις ε, κρίσεις είναι συμμετρικής φύσεως, οπότε όταν πλήττε κάποιος ε, πλήττονται και οι υπόλοιποι και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Να ξεκινήσω τις ερωτήσεις μου με την αρχή Τιμπεργκ την οποία ανέφερε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε πολλά εργαλεία, α, τόσα όσα και τα προβλήματά μας. Ίσως οι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε μια μακρόπνοη προσπάθεια ε, για τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, ίσως υποτιμούν ότι ένας από τους λόγους που έχουμε τόσα προβλήματα με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες είναι ότι ο σχεδιασμός ε, της ε, συνθήκης της, του Μάστριχτ και όλων των υπολείπων δεν έλαβε υπόψη τους, ε, τα μηδενικά κατώτερα επιτόκια. Επομένως κάτι μας λείπει. Μας λείπει ένα εργαλείο και στο βαθμό που δεν έχουμε αρκετά εργαλεία θα πρέπει να αρχίσουμε να στρεβλώνουμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη με τέτοιο τρόπο πια δεν θα μπορούμε να εξηγήσουμε τίποτα στον κόσμο. Εξού και τα προβλήματα που έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε και οι Υπουργοί Οικονομικών. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, πιστεύετε ότι το να δημιουργηθεί μια εύλογη δημοσιονομική ικανότητα θα μας βοηθήσει να πλουστεύσουμε τους κανόνες, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον να μπορούμε να εξηγούμε καλύτερα στον κόσμο αυτό που κάνουμε. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Συνδέεται με τις πολιτικές εκκίνησης. Ε, κανόνες ή διακριτική ευχέρεια. Το δούνου του στο, στο... Ε, στην έκθεση ανέφερε ε, το δανεισμό όπως το μηχανισμό, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ένα μικρό ε, προϋπολογισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια, άρα αλλαγέ στι συνθήκε. Ποιο από αυτού του τομεί θα πρέπει να μα προσχολήσει καταρχήν. σω χρειαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Και τρίτη ερώτηση είναι ο φόβο ότι θα έχουμε μία ένωση με χρηματοδοτικέ μεταφορέ. Φυσικά το θετικό είναι ότι αυτή η ένωση μα δίνει και μια ασφάλεια. Αλλά υπάρχει ε, και μια επιπλέον δυνατότητα, τα δημόσια αγαθά. Πιστεύετε ότι στην Ευρωζώνη ε, διάφορα θέματα ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν, παροχή δηλαδή κάποιων υπηρεσιών, κάποια δημόσια αγαθά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα η Ευρωζώνη. Ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κέλμερ. Ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Ε, τα μοντέλα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά η... το αποφασιστικό είναι ποια νούμερα κρύβονται από πίσω. Ακούστηκε ότι χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και επίσης ακούστηκε ότι δεν θέμε μία ένωση πληρωμών, μεταφορών. Αλλά τι θα είναι αν δεν είναι μία ένωση δημοσιονομικών μεταφορών. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε με αριθμούς τι ύψος θα έχει αυτή η δημοσιονομική ικανότητα. Διάβασα την πρόταση και μιλάει για 1 έως 7% του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν έχουμε τώρα έναν προϋπολογισμό 145 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι 1% του ΑΕΠ, σας ρωτώ, από πού θα προκύψουν αυτά τα λεφτά, από τον φορολογούμενο, από ποιες χώρες, με ποια κλίδα κατανομής, ποιος θα τα λαμβάνει. Ποιος θα αποφασίσει αυτά τα ζητήματα, για ποια έργα. Έχουμε πράγματι στην ε, Ευρώπη τόσο θαυμάσιους ανθρώπους που μπορούν να αποφασίσουν το τι χρειάζεται πού σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν εκδώσουμε μια τέτοια επιταγή εν λευκό και βεβαίως θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Αλλιώς είτε θα έχουμε φρούδες ελπίδες, θα δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες κάτι το οποίο θα είναι τραγικό δεδομένο του Brexit ή ακόμη χειρότερα να συνειδητοποιήσουν το τι συμβαίνει οι πολίτες όταν θα λάβουν το λογαριασμό. Είχαμε και τις εμπειρίες ε, με την ε, συνθήκη του Μάστριχτ. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε εντελώς τα πράγματα, να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και μετά να συζητήσουμε εάν συμφωνούμε με ένα τέτοιο προπολισμό ή όχι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πύρκο Ροένεν Λέρνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βεβαία ότι όλοι συμφωνούμε πως η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή δεν ε, είναι μια ζώνη με τις ε, καταλληλότερες πολιτικές για ε, την καταλληλότερη οικονομική και νομισματική ένωση και επίση πιστεύουμε ότι βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι η Ευρωζώνη. Είτε θα βγει προ μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση και προ μια πολιτική ένωση ή Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα πετήσουμε περισσότερη πειθαρχία στις αγορές. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία είμαστε πολύ επικριτικοί ε, στην περισσότερη ολοκλήρωση και στη Δημοσιονομική Ένωση. Και αμφισβητούμε κατά πόσο χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ήδη έχουμε αυξήσει την αλληλεγγύη με και νομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις προς τον ε, Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Έχω μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι η Ευρωζώνη με μια δημοσιονομική ικανότητα θα δώσει τη λύση στα προβλήματά σας, γιατί τα παρόντα κράτη-μέλη και μέχρι τώρα μεταφορές δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και δυστυχώς το έχουν νιώσει και στο πετσί τους και οι Έλληνες. Πόσο ρεαλιστικό πιστεύετε ότι είναι και άλλες χώρες να ε, εχωρίσουν δημοσιονομικές αποφάσεις από την εθνική τους κυριαρχία σε ένα υπερεθνικό σώμα. Και μια άλλη ερώτηση προς τον κύριο Ντάισελμπρον, τον πρόεδρο του Eurogroup. Πρόκειται να εξετάσετε κάποιες εναλλακτικές λύσεις αυτής της πολιτικής ολοκλήρωσης, μια πιο light ευρωζώνη ε, λειτουργικά ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποχώρηση ενό κράτου μέλου από την Ευρωζώνη, χωρί ταυτόχρονα να χρειάζεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επιθυμεί να παραμείνει σε αυτή. Ευχαριστώ. Ως και ο των Φιλελεύθερων από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και αυτό είμαι εγώ. Κύριε Υπουργή, οι παρεμβάσει σα. δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία σύγκληση. Αλλά βλέπουν, ε, διαφαίνονται και διάφορα σημεία επί των οποίων πρέπει να γίνει περισσότερη συζήτηση. Να υπενθυμίσω ότι όταν δημιουργήσαμε το ευρώ, ε, ρωτηθήκαμε θα του δώσουμε μια οικονομική διακυβέρνηση ε, ή θα έχουμε ε, ένα, απλώς κανόνες, ε, κανόνες ε, συνειδιοκτησίας. Και αυτό κάναμε με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι κανόνες ε, τους παραβαίνει κανείς, τους παραβιάζει κανείς, και αυτό συνέβη πολλές φορές, δεν υπήρξαν κυρώσεις. Και μπορούμε να πούμε σήμερα, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν κανόνες εξαιτία αυτού. Δεν υπάρχει ούτε καν κυβέρνηση, βέβαια, διακυβέρνηση. Όταν μιλήσαμε για το πρόβλημα του προϋπολογισμού, ε, τίθεται το θέμα της διακυβέρνησης Ευρωζώνης. Πάρα αυτά. Και όσοι από εσά πιστεύουν ότι δεν είναι και τόσο άσχημη ιδέα, είναι μια συζήτηση, είναι μια άποψη που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Γιατί η Ευρωζώνη δεν υλοποιεί τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας κώδικας ε, σύγκλησης και την ενθάρρυνση που θα πρέπει να, κάνουμε, να δώσουμε στα κράτη τα οποία κάνουν μια προσπάθεια για να συγκλίνουν. Πώς το βλέπετε αυτό, σας φαίνεται πιθανόν Δεύτερον, Ποιε είναι οι αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να εκχωρηθούν στην Ευρωζώνη. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τα κράτη-μέλη μπορούν να διαθέσουν στον προπολογισμό της Ευρωζώνης αυτό που τους κοστίζει σήμερα η άσκηση αυτής της αρμοδιότητας. Γίνεται αυτό. Έπειτα, υπάρχει ένα πρόβλημα με, την, με το κοινωνικό μας σύνολο. Οι, οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν σε εθνικό επίπεδο ο καθένας. σε ευρωπαϊκό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα της Ευρωζώνης, ας πούμε, στο εσωτερικό του οποίου οι κοινωνικοί εταίροι της Ευρωζώνης θα συνέρχονται ούτω ώστε να βγουν λιγάκι από την υπερβολική εθνική τους θεώρηση, ούτω ώστε να συμπληρώσουν αυτή την, αυτό το κίνημα που γίνεται προς μια βέλτιστη οικονομική και νομισματική ένωση. Ο σκιώδης εισηγητής της ΕΚΟΝ της ομάδας μου δεν είναι παρόν. Η κυρία Νηριάδα δεν είναι παρούσα. Δεν βλέπω κανέναν άλλον την ομάδα της επίσης. Ο Φαμπιο Ντεμάση. Α, ναι, ο Φαμπιο Ντεμάση. Ευχαριστώ. Ένας υπουργός μίλησε για τα μυστικά του καλού γάμου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση είπε ότι μπορεί να απέχουμε μόνο έναν κλειδονισμό από ένα πολύ άσχημο διαζύγιο. Ένα τέτοιο, ένας τέτοιος κλειδονισμός μπορεί να είναι η Ιταλική τραπεζική κρίση. Συμφωνώ πως η νομισματική πολιτική έχει εξοδετερωθεί από την λιτότητα, από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δεν είναι οι σωστές και έπληξαν την ιδιωτική ζήτηση. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τον Έλληνα Υπουργό εάν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος ε, αν συνδέσουμε τη δημοσιονομική ικανότητα με το ίδιο είδος ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ε, έχετε εμπειρία στην Ελλάδα θα έχουμε τελικά εξουδετέρωση του μακροοικονομικού αποτελέσματος το οποίο θέλουμε γιατί τελικά θα έχουμε μέτρα τα οποία θα μειώνουν την ιδιωτική ζήτηση και μήπως θα πρέπει να αποσυνδεθούν τα δύο ζητήματα. Δεύτερον, προς τον ε, Γάλλο Υπουργό Οικονομικών. Η Ευρωζώνη είναι πολύ ετερογενής και γνωρίζουμε πως μια μεγάλη ένωση οικονομικών μεταβάσεων δεν είναι δυνατή γιατί και από νομική και από πολιτική σκοπιά Μήπως θα ήταν σωστό να μειωθεί η ανάγκη για τέτοιες μεταφορές με το να στηρίξουμε μια πιο συμμετρική διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπου ξέρουμε ότι έχει φτάσει στα όρια η Γερμανία εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί έχουμε κάποια ελλείμματα στην Ισπανία και την Ιρλανδία ιδιωτικά. Όταν ξέσπασε η ευρωκρίση. Πώς θα ήταν αυτό το κατάλληλο μέσο για να δούμε και το θέμα του ιδιωτικού χρέους στην Ευρωζώνη. Τέλος, για την δημοσιονομική ικανότητα. Ναι, ένα ερώτημα προς όλους τους υπουργούς. Είστε διατεθειμένοι να σκεφτείτε με τρόπο καινοτόμο, να δώσετε τραπεζική άδεια στο μηχανισμό σταθερότητας ή να υπάρχει η δυνατότητα ενός χρυσού κανόνα των επενδύσεων, ε, να εξαιρεθούν οι επενδύσεις από τους κανόνες για το έλλειμμα, παραδείγματος χάρη. Τέλος, για τον Ιταλό Υπουργό, η Ιταλία έχει αρκετή δημοσιονομική ικανότητα να αντιμετωπίσει την τραπεζική κρίση που πλησιάζει. Σας ευχαριστώ. Για την ε, Γκουε, δεύτερη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν άκουσα που ε, δώσετε το λόγο πριν στη συνάδελφο. Δυστυχώ κολλείται, την αναπληρώνω εγώ. Είπε ο Υπουργό από τη Μάλτα ότι δύο χώρε, η Γερμανία και η Γαλλία, δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση του δημοσιονομικού έλλειμματο. Και τώρα του υπόλοιπου επιβάλλουμε κυρώσει για να μην ξανασεβεί αυτό. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πόρο απέχει από την έννοια τη δικαιοσύνη. Γιατί τι προωθούμε τελικά. Λέμε ότι ο πρώτο που καταστρατηγεί, που παραβιάζει, δεν πληρώνει, ο δεύτερο το κάνει. Οπότε κάποιο θα φροντίσει να είναι ο πρώτο που θα παραβιάσει μια συμφωνία γιατί θα την πληρώσει ο δεύτερο. Επίση, ε, εμεί ε, προτιμούμε την ενίσχυση ενός μοντέλου ευρωπαϊκών ε, φορολογικών εσόδων και η προώθηση μιας δημοσιονομικής, μιας δημοσιονομικής ικανότητας με αναδιαμετική ισχύ. Για παράδειγμα, με ένα φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών ή με φόρο στον άνθρακα. Επίσης, ε, να λαμβάνουμε υπόψη τη μέση οικονομική ικανότητα των, του πληθυσμού των κρατών μελών και τα χρηματοπιστωτικά μέσα να τα αφήσουμε σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και χωρίς ε, όρους προηγούμενους και προαπαιτούμενα. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Ντάισελμπλουμ, γιατί είστε ένας από τους πέντε προέδρους. Χρειάζονται μηχανισμοί φυσικά, αλλά δεν θα πρέπει κανένας να μένει πίσω. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μιας δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με αυτή τη γνώμη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Ερνέστ Μαραγκάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε διστάμενες απόψεις, αναμενόμενο άλλωστε. Και κατά τη γνώμη μου εκινούμε από ε, μια θετική πεποίθηση για την ανάγκη και την μάλιστα την επιτακτική ανάγκη του καθορισμού και της κοινή εφαρμογής αυτής της έννοιας της δημοσιονομικής ικανότητας ε, για τη σύγκληση, περισσότερη ε, σύγκληση και απορρόφηση ασυμμέτρων και συμμετρικών κρατασμών όπως προβλέπει και η έκθεση. Θα επικεντρωθώ σε δύο σαφείς ερωτήσεις που απευθύνονται περισσότερο από τους άλλους, τον κύριο Ντάισελμπλουμ. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα σύγκλησης, έχουμε ένα μηχανισμό και μια ε, ηλυμένη απόφαση διαδικασία για να αποφύγουμε τις ανισορροπίες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ξεκίνησε και λήφθη υπόψη δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων στην πατρίδα μου, την Ισπανία, λόγω υπέρμετρου δημόσιου ελλείμματος. Βέβαια, ουδέποτε μέχρι στιγμής έχω ακούσει, ούτε άκουσα ακόμα ότι θα ξεκινήσει τέτοια διαδικασία επιβολής κυρώσεων για ανισορροπίες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, γιατί έλλειμμα ε, τρεχουσών λογαριασμών πάνω από 6%. Γιατί αυτό αναφέρεται, αυτό κάνει η Γερμανία, η Ολλανδία και είναι πολύ σαφές. Γιατί δεν το... Ε, γιατί επιβάλλουμε κυρώσει για ένα είδος μόνο ανισορροπιών και όχι για τις υπόλοιπες. Δεύτερον, Μιλήσαμε για, το, για την ασφάλιση ανεργίας, για το Rainy Fund, για το Ταμείο Απρόβλεπτων Αναγκών. Γιατί να μην έχουμε και ένα ταμείο από, από μόνο δημόσιο χρέος με ε, ε επιστροφών μέσω τακτικών εισφορών των κρατών μελών και γιατί όχι και νέων ε, φορολογικών ε, ή δημοσιονομικών μέσων ευρωπαϊκού βεληνικούς. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ αυτού του τρίτου δρόμου που σα ανέφερα. Θα συμφωνούσατε με, το, με τη γνώμη αυτή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την οποία συμφωνούμε. Επίσης, ε, πιστεύετε ότι είναι συμβατή η δημοσιονομική ικανότητα με τη συνεχή μέχρι τώρα πρακτική της γενικευμένης δημοσιονομικής ικανότητας ε, που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως φορολογικό ντάμπινγκ. Πιστεύετε ότι είναι συμβατό να ανοίξουμε τη δυνατότητα της δημοσιονομικής ικανότητας όπως θα οφείλαμε με την πρακτική αυτή του φορολογικού ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έικχαουτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους 7 υπουργού που αντιμετώπισαν αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση. Ακούγοντας σας όλους, έχουμε την αίσθηση ότι συμφωνούμε επί των αρχών, ότι πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ικανότητα εν γέννη, αλλά κάποιοι από εσά λένε ναι, αλλά πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθούμε, ποιε είναι οι προτεραιότητε, τι πρέπει να κάνουμε πρώτα. Ε, νομίζω ότι ο Μαλτέζο ε, Υπουργό το είπαν και ο κύριο Ντάσιμπλουντ είπαν. Πρώτα σύγκληση και εν συνεχεία α συζητήσουμε τα, τα επόμενα εργαλεία, έτσι, συνοπτικά. Το είπαν. Κύριε Τσακαλώτο, ενδιαφέρον είναι αυτό που είπατε. Ε, είπατε ότι σε αυτή τη φάση με πολύ λίγες δυνατότητες νομισματικής πολιτικής, πολύ λίγες δυνατότητες ε, δημοσιονομικής πολιτικής, ε, όπου ε, ο επιμερισμός κινδύνου με τον ιδιωτικό τομέα είναι χαμηλός, ε, οποιοδήποτε σοκ υπάρχει, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κραδασμός υπάρχει, ε, που θα χτυπήσει στους μισθούς. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε κάνει μία αρκετά ενδελεχή συζήτηση. Γιατί ενώ συζητάμε ενδελεχώς, ε, στην πραγματικότητα τρέχουν και κάποια επίγοντα θέματα. Κύριε Ντάσιμπλιν, είπατε, ας ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση πρώτα. Αλλά μέχρι να έχουμε αυτό το ε, σύστημα ευρωπαϊκής ε, εγγύησης, μάλλον των ε, ευρωπαϊκών καταθέσεων, τι κάνουμε. Ε, εάν κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν θέλουμε όλο το βάρος να πέφτει στους μισθούς, θα πρέπει να συζητήσουμε με μια αίσθηση έτσι κατεπήγοντος. Κύριε Ντάισεπλουμ και κύριε Σικλούνα, θα ήθελα να μου πείτε ε, και εσείς ότι συναισθάνεστε ότι είναι κατεπίγουσα αυτή η συζήτηση. Και δεύτερο ερώτημα προς όλους τους υπουργού. Καλό είναι που κάνουμε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η συζήτηση. Αλλά το βασικό θέμα φυσικά είναι πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση σε εθνικά κοινοβούλια. Γιατί συμφωνώ με όλους σας ότι αν την κάνουμε αυτή η συζήτηση μόνο εδώ, θα αποτύχουμε. Το ερώτημά σας είναι λοιπόν Πώς μπορούμε αυτή τη συζήτηση να την περάσουμε στα εθνικά σας κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Μάρκο Βάλλη τώρα. Και θα εκπροσωπήσει τον Μάρκο Τζάνι. Έχει τέσσερα λεπτά. Έτσι, τέσσερα λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τους υπουργούς που ήρθαν εδώ σήμερα να μας μιλήσουν. Είμαι πεπισμένος ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης αυτή τη στιγμή αφού ανάκουγε αυτές τις 7 παρεμβάσεις των Υπουργών Οικονομικών, θα αμφέβαλε πάρα πολύ για την επιτυχία των ε, προσεχών συζητήσεων για το μέλλον του, της ΟΝΕ. Γιατί μοιάζει σαν να παρακάμπτεται το πρόβλημα. Θρησκευτικά το παρακάμπτεται το πρόβλημα. Κανένας από εσάς δεν εστιάζει στο πραγματικό πρόβλημα ε, που είναι η ουσία της ΟΝΕ. Το ευρώ. Ο κ. Γκραμένια είπε ότι δημιουργήσαμε μία ένωση μεταξύ 19 ε, οικονομιών και γίναμε προθύστεροι. Δημιουργήσαμε πράγματα που έπρεπε να δημιουργηθούν ε, μετά πρώτα. Δημιουργούν ανισορροπίες και δεν τις βλέπετε. Είναι το γερμανικό πλεόνασμα που είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη ανισορροπία από τα ελλείμματα που θα συζητήσετε αύριο. Επομένω, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό για αυτό το γερμανικό πλεόνασμα, θα πρέπει να, βάλουμε, να καθίσουμε τη Γερμανία ενώπιον των ευθυνών τη απέναντι στην ΟΝΕ. Να ναι. τη δείξουμε ότι μια οικονομία, τη στιγμή που έχουμε σταθερέ συναλλαγματικέ ισοτιμίε, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τα νομίσματα. Όπω είπε και ο κ. Παντοάν, τι κάνουμε, υποτιμούμε του μισθού. Και συμπιέσουμε του μισθού. Επομένω, ή θα βάλουμε τη Γερμανία ενώπιον των ευθυνών ή δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για ε, Οικονομική και Νοσηματική Ένωση. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθείτε εσείς. Υπάρχει μια σύστηση κατεπήγοντος στην ε, Ευρώπη. Το είπε και ο προλαλή σα. Και για μια φορά συμφωνώ μαζί του. Ή θα βρούμε μια λύση, ούτω ώστε να δει η Γερμανία τις ευθύνε τη και ίσως με αυτόν τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, ίσως αυτό το πλεόνασμα να χρησιμεύσει για να βοηθήσει και τις ε, περιοχές που βρίσκονται σε ύφεση στην Ευρωζώνη, γιατί εκεί σε αυτές τις περιοχές έχουμε τεράστιο πρόβλημα ε, ανεργίας. Μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Λέτε ότι η Ευρωζώνη είναι η περιοχή όπου έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Εγώ όμως ακούω ανθρώπους που λένε ε, δανείσατε στην ε, Ελλάδα για να πληρώσει την πραγματικότητα τι τους τόκους. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σήμερα. Ή θα πάμε προς μία κατεύθυνση κοινή λογικής και θα εστιάσουμε στο πρόβλημα του ευρώ και θα το επιλύσουμε, έτσι, με κάποιο τρόπο, ή αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για διάλυση αυτής της ζώνης και μάλιστα γρήγορα, πριν γίνει με άτακτο τρόπο. Ίσως θα πρέπει να γίνει με έφτακτο τρόπο. Ή θα συμφωνήσουμε λοιπόν σήμερα για να διαλύσουμε με συντεταγμένο τρόπο αυτή τη ζώνη ή θα βρούμε ένα δημοκρατικό μηχανισμό και έφτακτο για να επιτρέψουμε ε, σε ένα κράτος, όπως συνέβη ήδη, ας πούμε, με τον Brexit, ας πούμε, να φύγει, αλλά ένα, μια χώρα η οποία θα είναι μέσα στην Ευρωζώνη που θα θέλεις να φύγει. Γιατί θα υπάρξουν τέτοια δημοψηφίσματα που θα πούνε τέλος χρόνου, τέλος χρόνου σε αυτό το project, τέλος χρόνου σε αυτό το οικοδόμημα. Εσείς συζητάτε με θρησκευτική ευλάβη, εκεί τα ίδια και τα ίδια και ξεχνάτε, ενώ συζητάτε όλα αυτά τα θέματα, ξεχνάτε το πρόβλημα του ευρώ. Εγώ εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαι το θέμα τη ε, διακυβέρνηση και προσπάθησα έτσι με ταπεινό τρόπο να το βάλω το θέμα του ευρώ στη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να δουν το ευρώ ω πρόβλημα, αλλά και όμω πρέπει να το αναγνωρίσουμε ω τέτοιο. Διερωτώ με, αν κάποιο στη συνεδριά σα σήκωσε κάποιο το χεράκι του και είπε Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτά τα πράγματα τα ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με την οικονομία. Είναι βασικά, είναι στοιχειώδη, είναι πεδαριώδη. Και όμω κανένα δεν τα συζητάει. Σα καλώ να το κάνετε. Γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα. Το ευρώ. Σα ευχαριστώ. Δυστυχώ ε, δεν προλαβαίνουμε για διαδικασία κατστιά για υποβολή ερωτήσεων και ζητώ συγγνώμη από του υπόλοιπου συναδέλφου που δεν ήταν σκιώδει ηγητέ για να δικαιούνται να μιλήσουν. Α, συγγνώμη. Ξέχασα τον Ζερόλ Φάντεμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είδατε το τι συνέβη με τα φώτα. Ε, συμβολικό νομίζω όταν ένας οργανισμός ή ακόμα και ένα κτίριο είναι σε παρακμή ε, βγαίνει κάποιος στη σκηνή και φωνάζει σβήστε τα φώτα και αυτό συνέβη ε, Λοιπόν, θα κάνω λίγο τον γελοτοπιό τώρα. Στα Ολλανδικά. Λοιπόν, ακόμα δεν ε, ε, συνειδητοποιήσατε καλά-καλά το χτύπημα του Brexit. Έχουμε τώρα την τραπεζική κρίση της Ιταλίας και εδώ πέρα παριστάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα συνεχίζετε εσείς με κάποια αφηρημένα σχέδια, προχωράτε την ατζέντα σας και στην ημερήσια διάταξη αναφέρετε δημοσιονομική ικανότητα. Και συζητάτε σαν να είναι κάτι το εφικτό αυτό, σαν να μην ακούσατε την ήπια προειδοποίηση του Σλοβάκου Προέδρου ότι δεν είναι η στιγμή για να γίνουν αυτά τα πράγματα άμεσα. Πρέπει λίγο να ε, ηρεμήσετε, δηλαδή το να συζητάμε για δημοσιονομική ικανότητα για να σταθεροποιήσετε το ευρώ, είναι κάτι το τελείως εξωπραγματικό. Αφήστε το κανένα ε, εξάμεινο και δεν υπάρχει καμία δημοκρατική νομοποίηση για να προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν τα ευρώφυλα κόμματα να παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Ήμουν στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και αύριο θα παρουσιάσει ο κύριος Φερχόφστατ μια ένωση για περαιτέρω ενοποίηση και με αλλαγή της συνθήκης ε, και οργάνωση συνέλευσης ε, κανένα κράτος μέλος δεν θα στηρίξει αυτή τη στιγμή μια συνέλευση και δεν θα περάσει από κανένα δημοψήφισμα, εκτός αν θέλετε και άλλα Brexit exit μάλλον για την ε, ακρίβεια. Αν είστε λογικοί, νομίζω θα τα ξεχάσετε αυτά για λίγο. Μάλιστα. Θα ακούσουμε τώρα τους υπουργούς. Θα πρότεινα να τους δώσουμε το λόγο με την αντίστροφη σειρά από ό,τι προηγουμένως. Ε, σας αφήνω ελεύθερους, αλλά ξέρω ότι εσείς ε, πιέζετε να φύγετε σχετικά νωρίς. Οπότε από σας εξαρτάται πώς θα ρυθμίσετε το χρόνο ομιλίας σας. Ο κύριος Πέτερ Καζιμίρ. Ε, ότι προνόμιο. Ευχαριστώ. Γενικώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση το πώς μια τέτοια δημοσιονομική ικανότητα θα χρηματοδοτηθεί. Ε, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο της συζήτησης. Οπότε απλώς θα επαναλάβω ότι πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την ανάγκη δημιουργίας μιας δημοσιονομικής ικανότητας. Γιατί φαίνεται να διαφαίνεται κάποια συνένεση, εδώ τουλάχιστον μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Δεν θα κατονομάσω συγκεκριμένους ε, συναδέλφου που διαφωνούν. Θα πρέπει μετά να βρούμε τις λειτουργίες και, τη, και τα μέσα και χρηματοδότηση. Είναι το τελευταίο στάδιο της συζήτηση. Νομίζω αυτή είναι η σωστή σειρά. Εγώ προσωπικά θα μπορεί να ακουστώ ερετικός. Θα μπορούσα να είμαι ανοιχτό σε ένα τέτοιο είδος χρηματοδότησης, αλλά δεν θα συμφωνήσουν ίσως τα κράτη-μέλη. Ίσως ε, ε εθνικές συνεισφορές σε ένα νέο ευρωπαϊκό φόρο. Θα μπορούσε να είναι αυτό μια απάντηση, μια λύση. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσα να αναφέρω και την ομάδα του Μάριο Μόντι, που για μια δεκαετία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, της ανέβρεσης δηλαδή των πόρων και των μέσων για την χρηματοδότηση της δημοσιονομικής ικανότητας. Και επίσης αναφέρθηκαν οι πιθανές αλλαγές και το πώς θα τι θα κάνουμε τις επενδύσεις. Σήμερα το αναφέραμε, είμαστε στο δεύτερο πυλώνα των επενδύσεων και θα πρέπει να δούμε πώς θα άρουμε τα εμπόδια πρώτα που μας υπονομεύουν. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε το διοικητικό άκθος, τη γραφειοκρατία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της Eurostat, γιατί η λογοδοσία της Eurostat επίσης είναι μείζον ζήτημα. Θα, θα επιληφθούμε και αυτό το θέμα τους στους επόμενους μήνες. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ντάισελμπλουμ. Um, just like to pick up on... Θα αναφερθώ σε μερικές ερωτήσεις, δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες, θα χρειαζόταν ώρες. Ο κύριος Μουρεσάν ρώτησε ποιες διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις θα βοηθηθούν από αυτό το μέσο. Έχει δίκιο. Νομίζω πως πολλέ ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις ε, είναι θετικέ από μόνες τους. Άλλε αποδίδουν στον προπολογισμό θετικά. Εξαρτάται βεβαίω από τον σχεδιασμό. Κάποιες ε, άλλες είναι πολιτικά μη δημοφιλείς γιατί αφορούν κάποια κεκτημένα δικαιώματα ή κάποιες ομάδες ε, συμφερόντων που έχουν τώρα κάποια δικαιώματα και θα φύγουν. Αυτό το ζήτημα λοιπόν το οποίο είναι εξόχως ε, πολιτικό οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθηθεί από μια δημοσιονομική ικανότητα που θα στηρίζει χώρες στην διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει πριν από λίγα χρόνια, μια σύνδεση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, με μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Να υπάρξει μια σύνδεση. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Νομίζω θα μπορούσε να είναι ένας δρόμος ε, που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Οπότε μην νομίζετε ότι μπορούν να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μόνο αν υπάρχουν λεφτά για ξόδεμα. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Υπάρχουν πολλές εμπειρίες ε, αλλά βεβαίω εξαρτάται από τον σχεδιασμό και το είδος ε, των μεταρρυθμίσεων που θέλει κανείς. Για τον κύριο Φων Βάιστσακα, για το κύριο του ερώτημα, αν θα μας βοηθήσει αυτό το μέσο να απλοποιήσουμε τους κανόνες και να τους εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Μάλλον όχι, γιατί οποιοδήποτε μέσο αυτού του είδους, εφόσον ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, θα απαιτεί αυστηρούς κανόνες. Ποιος ε, είναι εντός και εκτός. Γιατί αν είναι να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μιας ε, ομάδας ανθρώπων, πρέπει, πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τα μέλη της ομάδας. Οπότε το ερώτημα είναι πότε δικαιούται κανείς τέτοια στήριξη, είτε είναι επίδομα ανεργία, είτε στήριξη στις επενδύσεις, ε, πότε δικαιούται κανείς αυτή τη στήριξη. Δεύτερον, τι απαιτούμε από μια χώρα πριν μπορεί παραδείγματος χάρη να ενταχθεί στο σύστημα επιδομάτων ανεργίας. Φαντάζομαι πως θα απαιτηθούν κάποια διαρθρωτικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανεργία. Οπότε θα υπάρχουν ε, δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, ταυτόχρονα. Οπότε το πώς θα οργανωθεί η ελληνική είναι θέμα δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε μόνο να παίρνουμε από το σύστημα, πρέπει και να εισφέρουμε είναι κάτι το απλό λοιπόν που θα εξηγείται απλώς, μάλλον όχι. Και έρχομαι άρα σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί εμένα ιδιαίτερα. Εάν γίνουν βήματα προς τα εμπρός και βρεθούν πολιτικοί συμβασμοί και βρούμε κάποιους κανόνες και έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις ή ξέρω εγώ, μείωση του κινδύνου με ε, κοινή ανάληψη του κινδύνου, θα βοηθούσε το να τηρούμε όλοι τους κανόνες και όχι στην πρώτη ευκαιρία να ξεκινάει μια συζήτηση για το αν είναι σωστοί οι κανόνες. Εντάξει, είμαι πάντα εγώ διατεθειμένο. πάρτε με τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα τη νύχτας ε, για να συζητήσουμε αν είναι σωστοί μηχανισμοί. Αλλά τη στιγμή που έχουμε κρίση ή ένα επίγον πρόβλημα, ο Μπα Άικχαουτ με ρώτησε για το τι θεωρώ κατεπήγον. Υπάρχουν επίγοντα προβλήματα στην Ευρωζώνη, αλλά όταν ακριβώς έχουμε επίγοντα προβλήματα δεν έχει νόημα κάθε φορά να αρχίζουμε να συζητάμε τους κανόνες. Α τους εφαρμόσουμε και για το μέλλον ναι, συζητήσουμε το εάν χρειάζεται επανασχεδιασμό το πλαίσιο. Γιατί έτσι δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτά τα μέσα και ακόμα σηκώνει πολλή συζήτηση το θέμα και αναλυτική δουλειά, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια εμπιστοσύνη ότι αν υποθέσουμε ότι καταλήγουμε σε κάποια συμφωνία, βλέπουμε κάποια προσθέμενη αξία και δημιουργούμε ένα πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι θα τηρηθούν τα υπεσχημένα. Γιατί έχει γίνει πλέον θεμελιώδες αυτό το ζήτημα και λυπούμε που το λέω έτσι, αλλά είναι το, το βασικό για μένα. Η εφαρμογή λοιπόν είναι βασικό θέμα για να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών. Αυτά. Τα λίγα. Τελειώσατε. Σκεφτόμουν πως δεν ε, είχατε τελειώσει, πως θέλετε να προσθέσετε και κάτι άλλο αυτά όσα είπατε. Ο κύριο Οι ανισορροπίες ε, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες, πιστεύω. Το, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις που αντιμετωπίζουν το θέμα του ηθικού κινδύνου είναι σαν να ζητάμε τον τρανό μετάστρα σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν κάποιες λύσεις με κάποιο στοιχείο ε, ηθικού κινδύνου, παραδείγματο χάρη το ενιαίο ε, ταμείο εξυγίανσης. Αν επιλύσουμε αυτό το θέμα, τότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Πάντα κατηγορούμε τη Γερμανία. Γιατί έχει πρόβλημα με τον ηθικό κίνδυνο. Αλλά και στη δική μου ταπεινή οικονομία. Και εμεί αισθανόμαστε το ίδιο. Σε ό,τι αφορά την ελληνική με τον Ευρωπαϊκό Οσμό ε, Σταθερότητας, εμείς ε, συνεισφέρουμε 3,3% του ΑΕΠΑ Είναι το υψηλότερο ποσοστό. Πώς να εξηγήσω στο λαό μου ότι θα πρέπει να δανειστεί σε, με υψηλότερο επιτόκιο για να δανείσει, ας πούμε, σε άλλες χώρες σε χαμηλότερα επιτόκια. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Είναι θέμα ποιότητας σε αντιδιαστολή με την ποσότητα. Πριν περάσουμε στην ξέβρεση περαιτέρων λύσεων, ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε ήδη. Η απογευματινή συζήτηση στο Συμβούλιο ακριβώ αυτή ήταν. Συζητούσαμε τις επενδύσεις και τους δικούς μας κανόνες που φημώνουν τις δημόσιες επενδύσεις. Οι κυβερνήσεις θέλουν να επενδύσουν περισσότερο, αλλά δεν μπορούν να. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσοί κανόνες. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το ισχύον σύστημα με τους κανονισμούς και τα λοιπά και να βασιστούμε σε αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι το θέμα ε, ανισορροπιών ανάμεσα στις πλεονασματικές και σε ελληματικές χώρες. Τα ελλείμματα των ελληματικών χωρών είναι τα πλεονάσματα των πλεονασματικών χωρών. Όμως, η όλη δομή, το όλο οικοδόμημα πιέζεται συνεχώ. Και ποιο πιέζεται κυρίω, οι ελληματικέ χώρε. Κανένα δεν μιλάει για τι πλεονασματικέ. Αλλά και αυτέ πρέπει να κάνουν αυτό που του αναλογεί. Γιατί σε οποιαδήποτε ζυγαριά, αν θέλει ε, το ένα κομμάτι να ανέβει, θα πρέπει και το, να κατέβει, το δεύτερο να κατέβει λιγάκι. Επομένω, υπάρχει τεράστιο περιθώριο για να σημειώσουμε πρόοδο στην Ευρωζώνη, χωρί να βρούμε υπερβολικές και πολύ εφάνταστες ε, λύσεις. Ευχαριστώ ο Πιέρ Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια θα πω μόνο. Καταρχήν, η... το θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας ε, είναι πολύ φιλόδοξο και χρειαζόμαστε φιλόδοξα σχέδια, αλλά όπως έδειξε και η συζήτηση εδώ, υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που καλύπτονται από τη δημοσιονομική ικανότητα που είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε σε όλα. Το καλύτερο είναι να βρούμε πού έχουμε αλληλεγγύη, πού έχουμε συγκλήσεις και κοινά σημεία. Και νομίζω ότι από τη συζήτηση και τα σχόλια φάνηκε ένα ευρύ φάσμα απόψεων και αποκλίνωση μερικέ φορέ απόψει για τι μπορούμε να κάνουμε με τη δημοσιονομική ικανότητα. Οπότε, πού μπορούμε να βρούμε τις, τα κοινά σημεία. Σε επίπεδο 19, γιατί έχουμε την Ευρωζώνη, αλλά α μην ξεχνούμε ότι είμαστε 28 χώρες μέλη και στο μέλλον μπορεί να μείνουμε 27. Οπότε εγώ θα έλεγα να βρούμε τέτοια θέματα. Για παράδειγμα, κοινού ενδιαφέροντο, όπω οι επενδύσει. Είχαμε τη σχετική συζήτηση το απόγευμα και αυτό το δρόμο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε γιατί χρειαζόμαστε του η Περισσότερε περισσοτερες ενίσχυση των όλε Οπότε ευρωπαϊκέ χώρε. μπορούσαμε να βρούμε και κοινού στόχου για να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Επίσης, η έκθεση των πέντε προέδρων μας δίνει πολλά, πολλές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το μέλλον. Και μια έχουμε και μαζί μας τον Γέρον Τάισεμπλο, που είναι ένας από τους προέδρους και πρόεδρος και του Eurogroup, κάνει πολύ αξιόλογο έργο στην προσπάθεια εφαρμογής κάποιων τμήματων της έκθεσης των πέντε προέδρων, που χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα είναι ε, αυτά που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα, χωρίς αλλαγή των συνθήκων, και το δεύτερο τμήμα που αφορούν ένα μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Α μην υποτιμούμε πόσο δύσκολη διαδικασία είναι η αναθεώρηση των συνθηκών. Α επικεντρωθούμε στα βραχυπρόθεσμα, να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε άμεσα με την αναζήτηση των κοινών σημείων και μια σταδιακή προσέγγιση και να εφαρμόσουμε μερικέ λίγε από τι ιδέε που υπάρχουν στο έγγραφο και που είναι πολύ φιλόδοξε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Πιερκάρλο Παντοάν. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα. Τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ε, χρειάζονται λεφτά για να εφαρμόσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όχι, αλλά βοηθάνε. Και Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πέρα από αυτούς που είπε ο Γερούν. Πρώτα απ' όλα είπαμε οι μεταρρυθμίσεις ε, αποδίδουν ε, μέσω αλλά τις πληρώνουμε εκ των προτέρων. Και δεύτερον, υπάρχουν περιπτώσεις όπως στη δική μου τη χώρα, όπου ο αντίκτυπος μεσοπρόθεσμα ενισχύεται από ένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό κίνητρο. Και αυτό σχετίζεται με τον ε, συνδυασμό της νέας εργατικής νομοθεσίας και των ε, επιδομάτων και των συμβάσεων ε, ορίστου χρόνου που θα αλλάξουν τη μορφή της αγοράς εργασίας. Δεύτερον, ο κύριος Τσέκερ αναφέρθηκε στο γιατί χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική ικανότητα. Ή ε, μίλησε για ευρωπαϊκά δημόσια καθά. Συμφωνώ πλήρω. Και έχω ένα παράδειγμα που νομίζω θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τη μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αποτελεσματική της μετανάστευσης απαιτεί την παροχή ευρωπαϊκών δημοσίων αγαθών που ορίζονται με διάφορους τρόπους αλλά εγώ σκέφτομαι ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τους, τους πρόσφυγες, την ένταξή τους στην οικονομία και παροχή πόρων για να μην βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή στις χώρες τους αφόρητη μέσα λοιπόν της βοήθειας των χωρών τους. Η παροχή λοιπόν ευρωπαϊκών δημοσίων αγαθών θα βοηθήσει τη συνοχή της Ευρώπης. Ένα παράδειγμα που νομίζω απαιτεί συλλογική δράση, η ικανότητα συλλογικής δράσης. Τρίτον, για την επαπειλούμενη τραπεζική κρίση στην Ιταλία που απαιτεί μεγάλη δημοσιονομική ικανότητα. Δεν υπάρχει τέτοια κρίση. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και θα πω αυτό το οποίο λέω και στον τύπο συνήθως. Τα νούμερα τα οποία ακούτε να κυκλοφορούν είναι απλά βλακίες. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα γιατί, αλλά μπορώ να σας δώσω τα πραγματικά νούμερα για το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι πολύ μικρότερο από αυτά τα οποία ακούγονται. Λίγες τράπεζες ε, έχουν πολύ υψηλό αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χρειάζονται χρόνο για να αντιμετωπιστούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί για να επιταχυνθεί η δικαστική πλευρά γιατί ξέρετε πως ε, αν μειωθεί ο χρόνος ε, επίλυσης ε, των διαφορών θα βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Δεύτερον, ο ιδιωτικό τομέα έχει φτιάξει κάποια συλλογικά μέσα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για τις ε, του ιδιωτικού τομέα, καθώς όπως ξέρετε δεν υπάρχει γενικώ η δυνατότητα να βοηθήσουμε με δημόσιο χρήμα λόγω κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Οπότε το θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραπεζών ε, είναι κάπως ε, εκτός θέματος. Και τέλος έχουμε ένα μέσο προφύλαξης ε, το οποίο συμφωνεί πλήρως με τους ε, κανόνες ε, περί δημοσίων ενισχύσεων για να αντιμετωπίσουμε πιθανώς κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια ευπάθεια. Αυτό για να ξεκαθαρίσουν διάφορες παρεξηγήσεις που κυκλοφορούν. Ευχαριστώ. Ο Ευκλής Τσακαλώτος, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Παλιά, δηλαδή δεκαετία του 90, πώς θεωρούν τα παιδιά μου. Εγώ θεωρώ ότι οι παλιές καλές μέρες είναι ο Ρόμπεν των Δασών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε μία άποψη συγκεκριμένη για τη σύγκληση και την αλληλεγγύα και το ίδιο συμφέρον. Ήταν τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό ήταν ο τρόπο που τα αντιμετώπιζε δεν ήταν απλώς ε, αλληλεγγύη, ήταν και ίδιο συμφέρον. Δηλαδή ότι εάν ο εταίρος μου δεν αναπτυχθεί, δεν θα είναι καλό για τις εξαγωγές μου. Για τις εξαγωγές μου. Το 2000 όμως άλλαξαν όλα αυτά. Ε, στην εφηλελεύθερη περίοδο αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε πια τα διαφορετικά ταμεία, αλλά μόνο στις ιδιωτικές ροές κεφαλαίων. Δηλαδή, τα λεφτά φεύγανε από τις πλούσιες χώρες, τις φτωχές χώρες, από τις ιδιωτικές τράπεζες, δημιουργούσε ζήτηση, για τα γερμανικά και ολλανδικά προϊόντα και αυτό το σύστημα λειτουργούσε μια χαρά. Υπήρχε θαυμάσια σύγκληση στη δεκαετία του 2000, αλλά το σύστημα κατέρευσε. Επομένω το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε την αντίστροφη πορεία. Δεν ισχύει ότι ο Βορρά απλώ δείχνει αλληλεγγύη, κερδίζει. Έχει πολύ χαμηλά επιτόκια. Και έχει ε, ροέ από τον Νότο στο Βορρά. Το αντίθετο από αυτό που η Ορθόδοξη Οικονομία λέει. Ε, Υποτίθεται ότι τα λεφτά ας πούμε, πηγαίνουν από τι φτωχέ, από τις πλούσιες Στην πραγματικότητα εδώ πέρα πηγαίνουν από τι φτωχέ στι πλούσιε. Οποιοδήποτε με ρωτάει, ε, ο Πιέρ πούμε, ο Σίγκριντ, ε, η κυρία από τη Φιλανδία με ρώτησε. Τι γίνεται με την αλληλεγγύη. Το πρώτο που πρέπει να αποφασίσουμε είναι αν έχουμε κοινό συμφέρον. Έχουμε κοινό συμφέρον όλοι μας να είμαστε καλά και ευημερούντες. Εάν δεν απαντήσουμε σωστά αυτό το ερώτημα, ε, τότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Με το ερώτημα αν έχουμε ένα κοινό συμφέρον, ε, να αναπτυχθούμε όλοι μας. Νομίζω ότι το μοντέλο της δεκαετίας του 2000 ε, ήταν λάθος, κατέρευσε. Θα πρέπει να έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο γιατί η ζήτηση είναι σημαντική και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ε, λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση. Γιατί ο κόσμος θέλει να κοινοτομήσει, να δεχτεί νέες κοινοτον... τεχνολογίες όταν δεν φοβάται για τη δουλειά του. Παίρνει ρίσκα όταν δεν φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. Επομένως, είναι σωστό αυτό. Επίσης, σημαντικό είναι να περάσουμε σε θετική ε, ενσωμάτωση. Οι αγορές δεν λύνουν από μόνες το πρόβλημα. Σε αυτά τα 8-10 χρόνια πριν την κρίση δεν έλυσαν το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε στοιχεία θετική ολοκλήρωση, να δημιουργήσουμε νέου δεσμού για την καινοτομία. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιε από τι ιδέε τη έκθεση και να τι υλοποιήσουμε και μόνο τότε. Και μόνο τότε, αν πάρουμε αυτές τις κοινέ αποφάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε. Το κοινό συμφέρον είναι προς το καλό όλων των Ευρωπαίων. Αν απαντήσουμε σε αυτό, έχει καλός. Αλλιώς, ας πάμε στο ανταγωνιστικό, στην ανταγωνιστική υποτίμηση, στις φυγόκεντρες τάσει. Η Γερμανία και η Ολλανδία θα έχουν ε, πολύ υψηλέ συναλλαγματικές ε, ισοτιμίες. Και ας πάμε από εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Επομένω, αν θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα χρειαζόμαστε περισσότερη ελληνική, το ερώτημα είναι καταρχάς που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν έχουμε κοινό μέλλον. Και μπορούμε να πάρουμε ιδέες από αυτή την έκθεση, από άλλες εκθέσεις και να προχωρήσουμε, βρίσκοντας μαζί λύσεις. Σας ευχαριστώ, Μισελ Σέπα. Ευχαριστώ. Είμαι τελευταίος, αλλά δεν φταίω εγώ για την καθυστέρηση. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Ο ευκλήδη έχει δίκιο. Στην ερώτηση έχουμε κοινό συμφέρον, η απάντηση είναι καταφατική. Δεν θα ήμουν εδώ, δεν θα ήμουν Ευρωπαίος, δεν θα ήμουν μαζί σας αν δεν συμφωνούσα ότι έχουμε κοινό συμφέρον ε, και συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση τα οικονομικά, δημοσιονομικά, νομισματικά θέματα. Όλα, συμμετέχουμε σε όλα αυτά για να προσπιστούμε το κοινό μα συμφέρον. Και αυτό που παλιά λέγαμε ευημερία, δυνατότητα ε, και η επόμενη γενιά να έχει λίγο περισσότερο και λίγο καλύτερη κατάσταση από τι προηγούμενε γενιέ. Αυτό, αυτό είναι το σχέδιο που θα πρέπει να μα εμπνέει όλου. Πληθώρα ήταν οι ερωτήσει που υποβλήθηκαν και μεγάλο το φάσμα και πολλές αποκλήσεις, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο-τρία πράγματα. Η αναζήτηση της δημοσιονομικής ικανότητας έρχεται σε αντίφαση με την ε, επιτυχία της νομισματικής πολιτικής. Όχι, η νομισματική πολιτική ήταν επιτυχής και το λέω ξεκάθαρα και ήμουν υπουργό Οικονομικών κατά τη συνθήκη της Μάστρικ και είδα όλη την εξέλιξη. Αλλά η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν αρκεί για να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων. Δεύτερον, η νομισματική πολιτική ή η δημοσιονομικη ικανότητα έρχεται σε αντίφαση με τις διαρθρωτικές πολιτικές. Όχι, οι διαρθρωτικές πολιτικές είναι και απαραίτητες, απολύτως απαραίτητες για τις χώρες και δεν δημοσιονομική πολιτική. Και μάλιστα σα προσκαλώ στη Γαλλία, γιατί και εδώ και σε εμά είναι δύσκολες οι μεταρρυθμίσει όπως όλες οι χώρες, αλλά γίνονται. Τρίτον, μας απαλλάσσει κάτι τέτοιο από την ε, ε, αναζήτηση συγκλήσεων και εφαρμογή συγκλήσεων σε θέματα δημοσιονομικά ή κοινωνικά. Όχι, δεν μας απαλλάσσει από κάτι τέτοιο. Γιατί χρειαζόμαστε και κάποιο του σύγκληση που δεν ε, θα επικεντρώνεται μόνο στα ωφέλη των διαρθρωτικών πολιτικών, αλλά θα εμπεριέχει και άλλες πολιτικές. Ή μας απαλλάσσει κάτι τέτοιο από την εμβάθυνση αυτού του σημαντικού ζεύγους της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μας, αν ε, κάθε χώρα που σέβεται αυτούς τους κανόνες ε, δεν δεν δείχνει την απαραίτητη ευθύνη, δεν αναλαμβάνει την απαραίτητη ευθύνη. Δεν νοείται αλληλεγγύη χωρί ευθύνη, χωρί υπευθυνότητα. Πρόκειται για ένα δίδυμο. Και μάλιστα η δημοσιονομική ικανότητα έρχεται ω κάτι επιπλέον, ω ένα συμπλήρωμα και κατά τη γνώμη μου απαραίτητο στοιχείο για να επιτύχουμε το κοινό μα σχέδιο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Τώρα κύριε Εισηγητρία, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργή. Δεν ξέρω που κρύψατε τις γυναίκες. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε και για αυτό το θέμα λύση. Με τον Ράιμα Μπέγκετ, τον οποίο θα ενημερώσω καταλεπτός για όλες αυτές τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψε, γιατί πραγματικά λυπάται που δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, δεν είμαστε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που έκανε μια έκθεση πρωτοβουλία ε, ω αυτό σκοπό για το θέμα τη δημοσιονομική ικανότητα Ευρωζώνη. Αλλά όλοι και οι εμπειρογνώμονε και οι ακαδημαϊκοί από τη στιγμή που άρχισαν να ασχολούνται με την ΟΝΕ άρχισαν να μιλούν και για την δημοσιονομική ικανότητα. Εκθέσεις Βέρνερ, Μακντούγκαλ, ε, Λονό, ακόμη και η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν είναι δική μας ιδιοτροπία ή δεν είχαμε τι να κάνουμε και κάναμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Εδώ και καιρό αναφέρεται αυτό το θέμα. Τώρα, έχουμε κάποια μέτρα ή εργαλεία σύγκλησης η έκθεση Delors, και σας παραπέμπω σε αυτή, έλεγε ότι από τη στιγμή που θα περάσουμε στο κοινό νόμισμα στο ευρώ, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία και να τα αναπροσαρμόσουμε στο κοινό νόμισμα. Βέβαια δεν ήμασταν όλοι στην Ευρωζώνη, όντως. Οπότε δημιουργήθηκε μια τελικά μια δημιουργική αμφισημία. Έχουμε ένα προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουμε προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Και έχουμε και κάποια διαρθρωτικά ταμεία που αφιταλαντεύονται μεταξύ των δύο. Και γι' αυτό και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και η Νομισματική μας Ένωση και η Νομισματική μας πολιτική διατρέχει κίνδυνο. Ε, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το δίπτυχο και το εξάπτυχο σύμφωνο. Και ότι όλα θα γίνουν καλά μετά, όλα θα πάνε καλά. Αλλά και τα δύο αυτά σύμφωνα, το δίπτυχο και το εξάπτυχο, είναι ε, ιδιώνησε ένα λάθος που ξεκινήσαμε, ότι έχουμε κανόνες που δεν εφαρμόζονται, άρα ε, χαλαρώνει η εμπιστοσύνη. Θέλουμε πιο αυστηρούς κανόνες για να ανακτήσουμε ή να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η συζήτηση που ξεκίνησε από την έναρξη του Συμφώνου Σταθερότητας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αντικειμενικά να κοιτάξουμε την κατάσταση σταθεροτητα και πιστευω οτι θα πρεπει αντικειμενικα να κοιταξουμε την κατασταση καταματα και να διαπιστώσουμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και άρα, από τη στιγμή που κάνουμε τη διαπίστωση ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Και νομίζω ότι μία από τις χρήσιμες και επικοδομητικές προτάσεις της έκθεσης πρωτοβουλίας μας και ελπίζω να την λάβετε υπόψη και να, πάρουμε, να πάμε και πιο πέρα από την έκθεση των πέντε προέδρων, προηγήθηκε του Βρετανικού Δημοψηφίσματος. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ιδέα του κώδικα σύγκλησης, την ανέφερε και ο πρόεδρος Αρτουή. Βλέπω ότι τα μεγάλα κατάμαυρα μάτια σας μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να βάλω τελεία. Λοιπόν, πίσω από αυτό το κώδικα σύγκλησης, τι βρίσκεται. Η αναζήτηση της ε, αρετής, ε, ε, όπως στην τη στιγμή που στην Ευρωζώνη είχαμε σύγκληση και από τη στιγμή που το κάναμε ήταν πριν το πέρασμα στο ευρώ, στο κοινό νόμισμα, γιατί τότε υπήρχε αποφασιστικότητα σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των κριτήριων του Μάστριχτ. Σας ευχαριστούμε κυρία Συνεισηγήτρια και ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους υπουργούς είναι σαφές ότι υπάρχει μια ταυτότητα και υπάρχει μια πραγματικότητα της Ευρωζώνης, γιατί τη στιγμή που χρειάστηκε, να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να συστήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής ε, Ασφάλειας, ε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αλληλεγγύη. Και ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμφαλαιότητά σας και την ηρεμία σα και την πρότητά σα, αλλά εμεί ω ε, ευρωβουλευτέ κρίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη συζήτηση τη Ευρωζώνης, τη διακυβέρνηση Ευρωζώνη και του προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Νομίζω ότι ήταν πολύ θαρρυντική αυτή η συζήτηση. Σα ευχαριστώ θερμά και να σα υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί, στη Βράση κολλάει το σίδερο, θα συνεδριάσουμε στις 11.30, 11.30 με 1, στην αίθουσα Γιάν 4Q2, για να εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, του σχεδίου έκθεσης και να προσπαθήσουμε να διαγράψουμε ίσως και τις, ε, να σχηματίσουμε τις αρχικές συμβαστικές